Ladies Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλώς ήρθατε <laughs> στην ε, σημερινή μας συνεδρίαση. Έχουμε πολλά διαφορετικά θέματα στην ημερησία διάταξη. Θα ξεκινήσουμε με ένα μεγάλο πακέτο, ε, τα θέματα 10, 11, 12, 13, τα οποία θα συζητήσουμε μαζί. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Ε, εισηγητής είναι ο, ο συνάδελφος Μπρεζίνα για όλα τα θέματα αυτά. Πολύ δουλειά σας περιμένει, ε, πολλά θέματα έχετε να εξετάσετε. Θα τα συζητήσουμε μαζί λοιπόν. Εάν συμφωνούν οι συνάδελφοι που είναι παρόντες, θα ξεκινήσει ο κύριος Μπρεζίνα την παρουσίασή του. Παρακαλώ. Uh, Κύριε Πρόεδρε, ε, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω ένα νομοθετικό πακέτο για το πρόγραμμα ε, πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ε, για το 2012-2013. Το νομοθετικό πακέτο αποτελείται από το πρόγραμμα πλαίσιο, συγκεκριμένα προγράμματα για το κοινό κέντρο ερευνών, καθώς και κανόνες για τη συμμετοχή. Η ε, συνθήκη Ευρατόμ περιορίζει τα προγράμματα στον ε, πυρηνικό τομέα ε, σε πέντε χρόνια. Τα ε, τα προγράμματα λήγουν το 2011. Γι' αυτό το νομοθετικό πακέτο στόχο έχει να στηρίξει ε, σύμφωνα με τις παρούσες νομοθετικές προοπτικές 2007-2013 ε, να στηρίξει λέω τις τα προγράμματα ατομικής ενέργειας. Για τους ε, συναδέρφους που παρακολουθούν τις εξελίξεις σε χώρες που έχουν αποφασίσει ε, την έξοδο από την πυρηνική ενέργεια, θα ήθελα να τονίσω ότι η νομοθεσία αυτή ε, ασχολείται μόνο με την έρευνα στον πυρηνικό τομέα και όχι με την οικονομική εκμετάλλευση της οικονομικής ενέργειας. Η καταστροφή της Φοκοσίμα θα πρέπει να μας δώσει κίνητρο να αυξήσουμε τις γνώσεις μας και την τεχνογνωσία μας στον τομέα αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε περισσότερη, όχι λιγότερη πυρηνική έρευνα που να έχει να κάνει και με την ε, ε, σύνδεξη ε, και θέματα όπως είναι η ασφάλεια, οι γιατρικές εφαρμογές και η ανάπτυξη νέων θεραπείων είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να συνεχιστούν. Τέλος, Είναι απαραίτητη η κοινή ευρωπαϊκή εκπαίδευση για να υπάρχει ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη ε, και ε, επιστημονική αριστεία και ανάπτυξη. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι όλα τα θέματα τα οποία ε, θα καλύπτονται από την ομοθέσια αυτή έχουν να κάνουν με την έρευνα και την ανάπτυξη και όχι με την οικονομική εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας. Ε, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας εδώ ο οποίος ε, επειδή ενδεχομένως ε, είναι κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για, παραγωγή ενέργειας να είναι κατά και των επιστημονικών προγραμμάτων. Άλλωστε οι προτάσεις Ευρατόμ συνδέονται στενά με άλλες δράσεις της Ένωσης όπως είναι το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 και οι στρατηγικές ενέργεια 2020. Ε, προσλέπω στην καλή συνεργασία με όλους τους συναδέρφους, σκιώδεις εισηγητές. Ε, είμαι ανοιχτός σε συζητήσεις και διατεθειμένος να βρω ε, συμβιβασμούς ώστε να μπορούμε να κάνουμε κάτι για τον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ που μας θυμήσατε ποιο είναι το θέμα μας ε, στην νομοθεσία αυτή. Ε, η κυρία Μαντουρέλ έχει ζητήσει πρώτη το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Χέρτσοφ που είναι σκιώδης συγγήτρια. Μου ζήτησε, μου έδωσε γραπτά την παρέμβασή της και θα σας την διαβάσω. Βέβαια τα έχει γράψει αγγλικά καλύτερα από τα δικά μου, αλλά θα σας έλεγε τα εξή. Ξέρουμε ότι τρέχουσες διατάξεις όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο της Euratom για την έρευνα και την κατάρτιση εκπνέει στο τέλος του 2011. Καθότι από τη συνθήκη προβλέπονται μόνο πενταετή προγράμματα. Οπότε έχουμε την πρόταση τώρα ε, του Συμβουλίου όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο για την περίοδο 2012-2013 και δύο επιπλέον προτάσεις απόφασης του Συμβουλίου που έχουν να κάνουν με άμεση και έμεση έρευνα στον ε, τομέα ειδικών προγραμμάτων. Συμφωνούμε για το πρόγραμμα πλαίσιο 2012-2013 στον τομέα της ε, έρευνας, ώστε να αναπτυχθεί έρευνα για ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια. Στον τομέα της ε, πυρηνικής ε, σύνδεξης, προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται καλύτερα τα ωφέλη από την ενέργεια στις ιατρικές επιστήμες, στην εκτινοβολία κτλ. Θέλουμε να αποφύγουμε βέβαια την ε, παράνομη χρήση, την παράνομη μεταφορά ενέργειας. Ήτρε λοιπόν συμφωνεί με τις ε, αρχικές πιστώσεις έτσι όπως προβλέπονται στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013. Αντιλαμβανόμαστε ότι το κόστος αυξάνει. Πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν με τα ποσά αυτά εφόσον θεωρείται εφικτό και μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα περιθώρια από άλλους τίτλους. Το ανώτατο ποσό για την εφαρμογή του προγράμματος πλαισίου, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, θα είναι 2,5 δισεκατομμύρια σε υποχρεώσεις. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί ως εξής. Για το ειδικό πρόγραμμα για έμεσες δράσεις, για την σύνδεξη και το ΙΤΕΡ, 2,2 δις, για την πυρηνική εισήδηξη και την προστασία από την ακτινοβολία 180 εκατομμύρια. Και, για το και προκειμένου το ειδικό πρόγραμμα να προχωρήσει για άμεση δράση, προβλέπονται 233 εκατομμύρια. Τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνουν και πρόταση για 100 εκατομμύρια 2012 και 160 το 2013 και υπάρχει και η νέα, πρόταση για να αυξηθούν τα ποσά του πολιτού ε, πλαισίου το 2012 στο 1α 650 εκατομμύρια για το 2012, λέμε, για το 2013 190 εκατομμύρια. Και τα δύο εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 20 Απριλίου του 2011. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση της Επιτροπής για το πολιετές ε, πρόγραμμα πλαίσιο, η αύξηση για το 1α με τις οροφές όσον αφορά το 2012 και το 2013 σημαίνει μείωση στο κεφάλαιο 2 και 5 κατά 240 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την εισηγήτρια δεν μπορούμε να αφήσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για το ίτερ. Πρέπει να βρει μια άλλη δημοσιονομική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό το θέμα τι θα κάνουμε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, λόγω της Φουκουσίμα, υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυρηνικά. Και γι' αυτό τίθεται το ερώτημα πώς στην εκπαίδευση μπορούμε να θέσουμε υψηλότερα πρότυπα. με συνεργασία, μέσω συνεργασίας με την ε, Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ε, ε, θα πρέπει να πετύχουμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στην Ευρώπη. Όσον αφορά την πυρηνική σύνδεξη, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε το πρόγραμμα βασικής έρευνας για τις νέες προτάσεις χρηματοδότησης. θα πρέπει να προβλέψουμε ειδική γραμμή για το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφος Τοσνόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη υπόθηκαν από τους προλαλήσαντες. Μπορώ να συμφωνήσω ε, σε πολλά σημεία με τον εισηγητή τον κύριο Μπρεζίνα και εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό να προχωρήσει η έρευνα στον τομέα αυτών και να υπάρξει σχετική χρηματοδότηση. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για ε, χρηματικούς πόρους που θα επενδυθούν ε, με πολύ χρήσιμο τρόπο διότι έτσι θα βελτιωθούν οι γνώσεις μας ε, και μάλιστα όχι μόνο στον πυρηνικό τομέα αλλά ε, και σε θέματα γιατρικής και άλλα. Νομίζω ότι πολλούς θα εξέπλητε αν συνειδητοποιούσαν πόσο ευρύ είναι το επίπεδο της ε, πυρηνικής έρευνας. Πρόκειται για, έρευνα, για επένδυση στο μέλλον μας. Ε, είναι κάτι που θα μας δώσει περισσότερες γνώσεις και που θα μας βοηθήσει σε πολλούς τομείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων μας. Επιπλέον, θεωρώ πολύ σημαντικό ε, το πρόγραμμα αυτό να καλύπτει και την εκπαίδευση. μετά από όλα τα προβλήματα που είδαμε μετά την καταστροφή στην ε, Φουκουσίμα, αλλά μετά και από την υπερβολική αντίδραση που είναι μεν κατανοητή, αλλά έχει οδηγήσει σε επιπλέον προβλήματα. τα γεγονότα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε παρανοήσεις και σε πολλούς άλλους τομείς. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντική αυτή η χρηματοδοτική πόρη. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε την κατάσταση μετά τη Φουκουσίμα, διότι φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν και σε τεχνικό και σε οργανωτικό επίπεδο. Αυτό φυσικά δεν ε, συνδέεται με το αν έχουν αποφασίσει κάποιες χώρες ε, να, ε, να ξεφύγουν από την ε, πυρηνική ενέργεια. Δεν θα πρέπει να χαθεί και η σχετική πυρηνική έρευνα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και δεν αφορά η έρευνα μόνο την παραγωγή ενέργειας. Σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση, διότι τα, οι έρευνες αυτές είναι πολύ ακριβές και μάλιστα ε, βρίσκονται σε έναν τομέα όπου είναι απαραίτητη η διεθνή συνεργασία, διότι πολύ λίγες χώρες έχουν ε, τη δυνατότητα τους πόρους ε, να κάνουν μόνες τους ε, τέτοιες έρευνες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προβλεφθεί και η ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των κέντρων. Τα προγράμματα αυτά είναι χρήσιμα, διότι έτσι αποφεύγεται και η επικάλυψη εργασιών. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τον κοινό στόχο. Είναι πολύ ε, καλή οι στόχοι που έχουν τεθεί και ως σκιώδης ε, εισηγητής ε, θα εργαστώ για να συμβάλλω στην ενέργεια αυτή, στην, στις προτάσεις αυτές, διότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν μπορούμε καν να γνωρίζουμε σήμερα τι σημασία θα έχουν αυτά τα θέματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο συνάδελφος Οντή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτή την δύσκολη υπόθεση. Έχω διάφορες παρατηρήσεις. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι το 2010 είχαμε αξιολόγηση αυτού του προγράμματος πλαίσιο. Εξάλλου είναι και υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αξιολόγηση αυτή πέρασε στα ψηλά ουσιαστικά. Νομίζω ότι ίσως τότε θα έπρεπε να είχαμε θέσει διάφορα ερωτήματα. Και προσθέτω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν κάνετε αξιολογήσεις, έγιναν καλά για το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά για την ε, Euratom νομίζω ότι η αξιολόγηση δεν ήταν ανεξάρτητη. Υπήρξε ένα πάνελ ανεξάρτητων ειδικών, αλλά πλαισιωνόταν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Και δεν νομίζω ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητο. Δεύτερον, οι προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προτάσεις οι οποίες συντάχτηκαν πριν από την τραγωδία της Ιαπωνίας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, η τραγωδία αυτή της Ιαπωνίας δεν πρέπει να οδηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σκεφτεί τι μηνύματα πρέπει να απευθύνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι έρχομαι τώρα στις παρατηρήσεις μου επί της ουσίας. Πρώτα απ' όλα για το ITER. Νομίζω ότι το είπαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα, οι σκιώδεις εισηγητές, ότι πρέπει να ε, δούμε την ε, αντίδρασή μας με στόχο την έρευνα. Ενώ στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάμε για οικοδόμηση. Νομίζω δηλαδή ότι την υποδομή της οικοδόμησης, από την οποία απορρέουν μεγάλα έξοδα φυσικά και πρέπει να το δούμε, αλλά πρέπει να δούμε και την έρευνα αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, χρηματοδοτούμε και προγράμματα έρευνας γιατί είχαμε πει ότι δεν θα χρηματοδοτήσουμε την εκμετάλλευση, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, αλλά προσοχή γιατί πρέπει να συγχρηματοδοτήσουμε και την έρευνα. Αλλιώς δεν πρόκειται να πετύχουμε πολιτική στήριξη. Όσον αφορά τώρα την κατανομή ανάμεσα στη σύνδεξη και στη σχάση. Η τραγωδία της Ιαπωνίας πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε περισσότερο και ρωτάω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ανοιχτή σε αυτό το ζήτημα Μήπως θα έπρεπε να έχουμε προγράμματα ερευνητικά, για παράδειγμα για τον παροπλισμό πυρηνικών εργοστασίων που λειτουργούν βάσει της τεχνολογίας χάσης. Τι εννοώ, ότι τα κράτη-μέλη σήμερα είναι κυρίαρχα όσον αφορά την ενέργεια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 50, σε 100, 150 χρόνια. Μιλάμε για παροπλισμό πυρηνικών εργοστασίων. Έχουμε εμείς οι Ευρωπαίοι τους καλύτερους μηχανικούς, την καλύτερη τεχνολογία για τον παροπλισμό τέτοιων εγκαταστάσεων. Είμαστε λοιπόν μπροστά και αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε. Γιατί έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και να τους διασφαλίσουμε ότι ό,τι ε, ε, ατομικές εγκαταστάσεις ε, έχουμε είναι τέτοιες που είναι καλυμμένες στην περίπτωση παροπλισμού με το σωστό κόστος και με τις καλύτερες προδιαγραφές. Και σίγουρα βάσει των προδιαγραφών έτσι όπως αυτές θα εξελιχθούν. Έχουμε προγράμματα για την τεχνολογία παραπλησμού. Δεν παροπλίζουμε ένα κινητήρα ε, ατομικού αντιδραστήρα με τον ίδιο τρόπο όπως το κάνουμε για έναν οποιοδήποτε άλλο κινητήρα. Για την κατάρτιση τώρα πρέπει να καταγράψουμε όλες τις σχολές ε, που έχουμε και απασχολούνται με αυτό το θέμα. Μετά το ατύχημα ε, στη Φουκουσίμα έχουμε διαπιστώσει ότι τελικά δεν έχουμε αρκετούς επιστήμονες ειδικευμένου σε τέτοια θέματα. Η διαχείριση της πυρηνικής ενέργειας, ο παροπλισμός ενός πυρηνικού αντιδραστήρα και αφορά όλες τις χώρες. Δεν υπάρχει μόνο το του στη Βουλγαρία, η Γερμανία και η Γαλλία θα αλλάξει γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων. Συνεπώς, έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Και από την άλλη μεριά, όταν βάζουμε πολλά χρήματα στο ίτερ, δεν ξέρω είναι άλλο θέμα, αλλά θέλω και αυτό να το θέσω, μήπως πρέπει να ξαναδούμε με τους εταίρους μας εκτός Ευρώπης ε, οικονομικές διαπραγματεύσεις. Και υπενθυμίζω ότι εμείς γνωμοδοτούμε. Εγώ είμαι από τους ευρωβουλευτές που εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι η Euratom δεν έχει κοινοβουλευτική διάσταση. Ευχαριστούμε κύριο Ζαντό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά για μένα να παίρνω το λόγο μετά από τον συνάδελφο Οντί δεν συμφωνούμε πάντα, δεν έχουμε πάντα την ίδια οπτική γωνία ή δεν προβάλλουμε στο μέλλον με τον ίδιο τρόπο τα πυρηνικά, ούτε όσον αφορά τη Γαλλία, ούτε όσον αφορά τον κόσμο ολόκληρο. Εσείς μιλάτε για 100-150 χρόνια, μιλάτε για άλλες γενιές πυρηνικών αντιδραστήρων. Θα δούμε. Θα δούμε ποιο θα είναι το μέλλον. Εγώ νομίζω ότι η οικοδόμηση νέων πυρηνικών αντιδραστήρων είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζετε εσείς στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Συμφωνώ όμω με του προλαλήσαντε για το εξή. Πρώτον, για το θέμα του παροπλισμού. Ναι, πράγματι, πρέπει να τίθεται το θέμα του παροπλισμού και να υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης για παροπλισμό. Ξέρουμε σήμερα, για όποια χώρα και αν πρόκειται, ότι δεν έχουμε αρκετούς μηχανικούς ειδικευμένου στον τομέα της ατομικής ενέργεια. Φεύγουν, βγαίνουν από την αγορά αυτοί που φτιάξανε τους ε, πυρηνικούς αντιδραστήριους που έχουμε σήμερα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα υπεργολαβίας με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι όπως θα έπρεπε για την ευαισθη... ευαισθησία ε, που περιβάλλει το θέμα της ατομικής ενέργειας. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να προσλάβουμε προσωπικό, μηχανικούς, ειδικευμένους στην ατομική ενέργεια. Και αυτό για να μπορούμε να τα βγάλουμε καλύτερα πέρα και για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο και όχι να δημιουργούμε ψευδεστήσεις ότι εγκαταλείπουμε τα πυρηνικά. Τώρα, για ορισμένου υπάρχει ιδέα ότι πρέπει να συνεχίσουμε ό,τι κάναμε και όπως κάναμε μέχρι τώρα, χωρίς να πάρουμε μαθήματα από τη Φουκουσίμα. Όμω, πριν από τη Φουκουσίμα, έτσι κι αλλιώς είχαμε μεγάλε αβεβαιότητες... για προγράμματα όπως το ITER όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους, τι ξέρουμε για μετά το 2013, μεγάλες αβεβαιότητες δηλαδή. Τώρα μετά τη Φουκουσίμα έχουμε νέες αβεβαιότητες για τις προθεσμίες και για το κόστος. Αβεβαιότητες που μας κάνουν να ξαναβλέπουμε τους στόχους μας για την ενεργειακή μας πολιτική. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αποσυνδέσουμε πλήρως την έρευνα από την ενεργειακή πραγματικότητα. Γιατί δεν είναι δυνατόν το κοινοβούλιο αυτό να επικυρώνει την ιδέα που λέει ότι ο προπολογισμό για τα, την ενέργεια φαίνεται σε, για τα πυρηνικά θα είναι 4,5 φορέ παραπάνω από ό,τι για τι αναλλακτικές ενέργειε. Μα αυτό θέλουμε, έτσι θέλουμε το ενεργειακό μα μέλλον στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Συνεπώ, όσον αφορά τον ερευνητικό προπολογισμό, ναι, να προσανατολιστεί προς τον παροπλισμό. Συμφωνώ και με τις ιατρικέ εφαρμογές, ασφαλώ. Αλλά όσον αφορά το ΙΤΕΡ, που είναι το μεγάλο κομμάτι, καιρό είναι να σταματήσουμε να ψάχνουμε, αλλά να δούμε με ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε προς τους ε, στόχους μας και να αποφασίσουμε μήπως πρέπει να σταματήσει ή μήπως πρέπει να προσανατολιστεί αλλιώς. Ίσως να αδράξω την ευκαιρία για να ρωτήσουμε την γραμματεία. Μας είπατε ότι πρέπει να μάθουμε από τη Φουκουσίμα. Το θέμα της πολιτικής, της πολιτικής αξιολόγησης έχει οδηγήσει σε διαφορετικές πολιτικές θέσεις, αλλά ένα θέμα είναι ενδιαφέρον το οποίο δεν έχουμε συζητήσει ποτέ. Ποτέ ε, δεν έχουμε εξετάσει τι ακριβώς ε, έγινε στη Φουκουσίμα. Ίσως θα ήταν χρήσιμο ε, σε κάποια από τις ε, επόμενες συνεδριάσεις, τώρα που έχει περάσει κάποιος χρόνος, που έχει μεσολαβήσει κάποιο διάστημα και που ίσως να γνωρίζουμε περισσότερο, ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιον να μας ενημερώσει. Ε, στο ζητώ λοιπόν από τη γραμματεία, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Χένεν. Ο κύριος Σανά. Λέμε στη Γαλλία ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σκεφτόμαστε λογικά. Η καταστροφή της Φουκουσίμα αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι κάθε βιομηχανική διαδικασία παραγωγής ενέργειας περιέχει κινδύνους. Και το άτομο ακόμα περισσότερο. Δεν μπορούμε ε, να καταλήξουμε σε πορίσματα, γιατί δεν έχουμε ούτε το 1 δέκατο των απαραίτητων ε, στοιχείων για να κάνουμε μια αντικειμενική ανάλυση της κατάστασης. Επίσης είδαμε ότι το γεγονός ότι είναι, πρόκειται για έναν ε, ιδιωτικό φορέα, ο οποίος διαρκώς προσπαθεί να μειώσει το κόστος για να υλοποιήσει όσο γίνεται περισσότερα κέρδη, σίγουρα αυτό δεν είναι η καλύτερη λύση και αυτό προκαλεί δυσκολίες για τους πολίτες που βρίσκονται γύρω εκεί και που εργάζονται εκεί πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η πρόταση να συνεχιστεί η έρευνα με ευφυΐα σε όλους τους τομείς για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των μισθωτών, των πολιτών, αλλά να εγγυηθούμε επίσης τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν μια θεμητή και οικονομική πρόσβαση στην ενέργεια είναι απαραίτητο. Εάν δεν το σκεφτούμε σήμερα, αν δεν δουλέψουμε σήμερα για να οικοδομήσουμε, να φτιάξουμε τις αυριανές ενέργειες, είτε είναι βιώσιμες, ανανεώσιμες, είτε και ατομικές, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε όλοι σήμερα, δεν θα τα καταφέρουμε και θα μείνουμε πίσω. Η κατάρτιση όλων των μηχανικών και όλων των τεχνικών που δουλεύουν στο σύνολο της ε, ενεργειακής διαδικασίας της ατομικής είναι απαραίτητη και πιστεύω επίσης ότι οφείλουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσουμε διάφορες ε, ε, παρατηρήσεις γιατί υπάρχει η υπεργολαβία της υπεργολαβίας στις πυρηνικούς σταθμούς η υπεργολαβία δίνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία κατάρτιση. Δίνεται στις φθηνότερες συντε... ε... ε επιχειρήσεις interim. Δεν συνέβη αυτό στη Φουκουσίμα, αλλά λέω ότι γίνονται πράγματα απαράδεκτα. Δεν μπορεί δηλαδή οι πολίτες να εξαρτώνται από τα 20, ευρώ, 20 λεπτά του ευρώ εξοικονόμησης για κάθε μισθωτό. Ε, έρευνα και για τις ανανεώσιμες. Όλοι ξέρουμε πώς προχωρούμε προς ένα μείγμα, ακόμα και αν έχουμε διαφορές για την πυρηνική ενέργεια. Είναι αλήθεια και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Η ε, Γερμανία κάνει μια ανακοίνωση ότι θα, σταματήσει την ατομική ενέργεια Μα θα αγοράσει από την Ιταλία, από τη Γαλλία. Η Ιταλία κάνει το ίδιο, μα θα αγοράσει ενέργεια από εμά. Εγώ προτείνω η Τσεχία και η Γαλλία να διπλασιάσουν το κόστος. Να διπλασιάσουμε την τιμή του, της ενέργειας. Αφού υπάρχει ζήτηση και δεν υπάρχει προσφορά, είναι η νόμη της αγοράς. Ε, ε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και να συνεχίσουμε να προχωρούμε ήρεμα. Οι πολίτες μας έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια, στην υγεία, στην κυριότητα του ω άτομα και έχουν και καθήκοντα. Να συμμετέχουν δηλαδή στην οικοδόμηση μια κοινωνία όπου καθένα έχει τι ίδιε δυνατότητε να τα καταφέρει. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο εμεί να βοηθήσουμε και να συνοδεύσουμε την κατάρτιση. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να σταματήσουμε, μην ξεχνάμε διαρκώς τα πράγματα. Είμαστε έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε αγωγούς φυσικού αερίου που θα περνάνε όλη την Ευρώπη και που θα εξυπηρετήσουν μεγάλους ομίλους που βάζουν ε, τα κέρδη τους σε λογαριασμού στην Ελβετία και τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και δεν θέλουμε να προχωρήσουμε και να στηρίξουμε αυτούς που δουλεύουν στους ατομικούς σταθμούς και παράχουν ηλεκτρισμό. Ας είμαστε σε θέση να δούμε ότι έχουμε ανάγκες για τον πληθυσμό μας και για τη βιομηχανία μας, αλλά ότι έχουμε και καθήκοντα να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την κατάρτιση των εργαζομένων. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ναι. Να προσθέσω κάτι. Ο συνάδελφος Πρεζίνα έφερε αντίρρηση όταν είπατε ότι οι Γερμανοί και οι ε, ε, Σλοβακοί θα πρέπει να ε, αγοράσουν την ενέργεια στην Γαλλία. Μας υποδεικνύει ότι υπάρχει και μια πρόταση της Τσεχίας, μια προσφορά της Τσεχίας, απλά για να είναι πλήρης οι πληροφορίες μας. Ο συνάδελφος Ρεμέκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε ότι κάποιες επιχειρήσεις ετοιμάζονται στην, να ε, ανταποκριθούν στην ε, απόφαση της Γερμανίας ε, να εγκαταλείψει την πυρηνική ενέργεια. Περιμένουν ότι οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν κατά 20%. Δεν ήταν αυτό όμως το σημαντικό που ήθελα να πω. Ήθελα να πω ε, αυτά που ήδη υπόθηκαν. Ε, θα χαρώ πολύ με την, ε, να συνεργαστώ με τον εισηγητή. Ο κύριος Μπρεζίνα είναι ειδικό σε τέτοια θέματα και είμαι βέβαιος ότι θα διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα στις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να τονίσω κάποιες πτυχές. Μιλάμε για εκπαίδευση, για έρευνα σε έναν πολύ ευαίσθητο τομέα. Μιλάμε και για μετεκπαίδευση και για επαγγελματική κατάρτιση. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μια σύγκριση με το παρελθόν. Ε, συνάδελφοι, ε, φανταστείτε ένα αεροπλάνο που πετάει ε, να σταματήσει η μία μηχανή, το προσωπικό, ο πιλότος προσπαθεί να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροπλάνο και εξετάζει κανείς εκ των υστέρων ε, γιατί δεν ε, λειτουργήσε ε, το τρίτο μοτέρ. Αυτό όμως δεν μπορεί να εξεταστεί κατά τη διάρκεια της πτήσης, πρέπει να γίνει μετά. Τώρα μετά την Φουκουσίμα συμπεριφερόμαστε σαν τους επιβάτες σε ένα τέτοιο αεροπλάνο που έχει πάθει βλάβη στο παρελθόν. Και λόγω της πράσινης πολιτικής ε, έχουμε επιφέρει μεγάλη ανασφάλεια στον τομέα αυτών. Οι εργαζόμενοι στον πυρηνικό τομέα έχουν αναζητήσει άλλες θέσεις εργασίας. Ο συνάδελφος Ενένα έχει δίκιο. Πάντα υπάρχουν ε, τεχνικοί κίνδυνοι και γι' αυτό θα πρέπει να στείλουμε ένα σημαντικό θετικό μήνυμα ότι είναι σημαντική η εκπαίδευση Και σημαντικό είναι ε, οι άνθρωποι του τομέα πάντα να μπορούν να βρουν δουλειά. Οι πολιτικοί ε, βρίσκονται στα χέρια των ε, εξειδικευμένων αυτών ανθρώπων που μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για την επίλυση περιπτώσεων ανάγκης. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, για τόσα όσα είπατε πριν από λίγο Όσον αφορά να ακούσουμε από κάποιον ε, με λεπτομέρειες την διαδοχή των γεγονότων στη Βοκουσίμα, δηλαδή τι ακριβώς συνέβη, την περασμένη εβδομάδα στη συζήτηση εγώ σας παρέθεσα από το σχέδιο έκθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την επιθεώρηση πυρηνικής ασφάλειας. τον επικεφαλής αυτής της υπηρεσίας και ξέρετε ότι αυτό έχει διοριστεί επικεφαλής της IAEA, e του Διεθνούς Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας, για να διερευνήσει ακριβώς τι συνέβη στη Φουκουσίμα. Θα μπορούσαμε να τον καλέσουμε εδώ και να ξέρουμε, να ακούσουμε ακριβώς τι συνέβη και την ανάλυση του. Να τον καλέσουμε για να παρακολουθήσει την Επιτροπή και να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση των πορισμάτων του. Επίσης, αυτό που λέτε ότι η πυρηνική ενέργεια είναι πιο επικίνδυνη από όλες τις άλλες, οι στατιστικές λένε άλλα πάντως. Λένε ότι ο αριθμός ατυχημάτων και απολειών ζωών σε άλλους ε, τομείς της ενέργειας ή στην εξόριξη πετρελαίου είτε στην υδροηλεκτρική ενέργεια και ιδιαίτερα στην εξόριξη άνθρακα ε, τα στοιχεία λοιπόν είναι πολύ πολύ χειρότερα από ότι αυτά στην πυρηνική, πολιτική πυρηνική βιομηχανία. Ξέρω βέβαια ότι ο κόσμος αντιδρά έντονα στις λέξεις «πυρνική ενέργεια. Αλλά ας μην μας κάνει αυτό να ξεχνάμε τα στοιχεία. Τα στοιχεία για την ασφάλεια της πυρνικής ενέργειας. Και τέλος, τρίτο σημείο με, σε σχέση με το τι θα συμβεί στη Γερμανία όταν θα σβήσουν οι προβολείς που φωτίζουν αυτή τη στιγμή την πυρνική ενέργεια θα σβήσουν οι προβολή σε καμιά δεκαριά χρόνια αφού δεν θα έχει πυρηνική ενέργεια πια η Γερμανία και ελπίζουμε ότι τότε μια νέα γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων θα αρχίσει να λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και ίσως θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε μέσω της δυσύνδεσης που περνά από το καράλι της μάχης. Ελπίζω τουλάχιστον γιατί διαφορετικά θα υπάρχουν πολλές διακοπές στην παροχή ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, τρίτη προσφορά ακούσαμε, πάρα πολύ ωραία. Θα προσπαθήσουμε να τη συγκεντρώσουμε όλες. Ε, ο συνάδελφος Ρίμπιχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα, παλά, ήθελα απλά να αναφερθώ στην δυνατότητα να λάβουμε πιο αναλυτικές ε, πληροφορίες σχετικά με την Φουκουσίμα. Ε, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα έναν εμπειρογνώμονα από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο, ο οποίος ε, μας ε, είπε ποια ήταν τα προβλήματα και ποιες ήταν οι συνέπειες. Θα πρότεινα λοιπόν να προσκαλέσουμε κάποιον από το Joint Research Center, το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο. Επίσης αναφέρθηκε στις οικονομικές συνέπειες αυτής της καταστροφής. Ε, θα φροντίσω στον ε, πρόεδρο να υποβάλω τα έγγραφα που μας ε, δόθηκε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση αυτή. Νομίζω ότι πολύ ευχαριστώ θα την υιοθετήσουμε. Ο κύριος Στασνόσκη. Συγγνώμη που ξαναπαίρνω το λόγο, αλλά Είμαι και εγώ υπέρ αυτή τη πρόταση. Ε, πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε μια τέτοια παρουσίαση. Συμφωνώ με όλου ε, του συναδέλφου που είπαν ότι θα πρέπει να προσκαλέσουμε ανθρώπου που είδαν πραγματικά τι έγινε ε, επί τόπου, ώστε να μην λάβουμε μόνο έμεσε πληροφορίε. Οι έμεσε πληροφορίε διαβρώνονται επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι η γραμματεία θα μπορούσε ενδεχομένω να σκεφτεί το εξή. Ε, η Ευρώπη έστειλε μία ομάδα διάσωσης ε, που αποτελεί το από ε, εμπειρογνώμονους σε, περίπτωση, σε περιπτώσεις τέτοιων καταστροφών, αλλά στάρισαν και οι ειδικοί του πυρηνικού τομέα. και ξέρω ότι βρέθηκαν πολύ κοντά στον τόπο της καταστροφής ε, και βοήθησαν ε, ε, στην στην διάσωση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα μπορούσαν να μας περιγράψουν τι ακριβως συνεβη συνέβη. Βρέθηκαν εκεί δύο-τρει εβδομάδες μετά την καταστροφή. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να σκεφτούμε μήπω θέλουμε να προσκαλέσουμε τέτοιου ανθρώπου στην παρουσίαση. Γενικά είμαι υπέρ τη οργάνωσης μιας μήνυα ακρόασης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συνάδελφος Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αυτό. Θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους από τα άλλα κράτη-μέλη που ε, προσφέρθηκαν ε, να μας προμηθεύσουν ηλεκτρική ενέργεια όταν δεν θα έχουμε πια στη Γερμανία. Ας δούμε τι θα γίνει. Άλλωστε δεν ε, θα έχουμε άμεση έξω από την πυρηνική ενέργεια, θα έχουμε βαθμιαία ε, κατάργηση. Ε, εδώ και χρόνια προσπαθούμε μάταια να οργανώσουμε την εσωτερική αγορά ενέργειας. Ας δούμε λοιπόν τι θα γίνει όταν εφαρμοστεί τελικά αυτή και άλλωστε ο ανταγωνισμός είναι καλός. Ε, προτείνω στους συναδέλφους τώρα που ε, σκιαγραφούν σενάρια τρόμου να, σκεφτούν, να εξετάσουν την ε, έκθεση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις αυτές. Ο συνάδελφος Οντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πολύ σύντομα. Είναι πολύ καλό να έχουμε εδώ το Κοινό Κέντρο Ερευνών που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε την δουλειά της Euratom. Συμφωνώ και στηρίζω την πρόταση αυτή. Ο κύριο Ζαντό. Μία πληροφορία θέλω να δώσω. Συμφωνώ και επικαιρώνω αυτά που είπε ο συνάδελφος. Οι Γερμανοί έχουν κάποιο λόγο. Εγώ ακούω ότι οι Γερμανοί ακούνε τον κόσμο στη δημοκρατία. Κάποιος σου μίλησε για φουλ, το πλήθος. Ε, δεν είναι έτσι. Πρέπει να χρησιμοποιούμε όρους στη δημοκρατία πιο ε, σοβαρούς για τον κόσμο. Αντί λοιπόν να ακούμε τα επιχειρήματα της πυρηνικής βιομηχανίας, σας κοιτάμε τις στατιστικές. Από τότε που έκλεισαν 7 και 1 αντιδραστήρες στη Γερμανία, ας δούμε τα στατιστικά στοιχεία τι γίνεται μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας με την ηλεκτρική ενέργεια. Όλα αυτά που λέει η γαλλική πυρηνική βιομηχανία και που τροφοδοτούν την Γερμανία δεν είναι αλήθεια. Επιπλέον, πρέπει να γίνει εξολόγηση του Φουκουσίμα. Ο συνάδελφος των ε, Πρασίνων, ο Μισελ είναι τώρα στην ε, Φουκουσίμα. Είναι η συγγήτρια για το θέμα αυτό και περιμένω να γυρίσει και να τη ζητήσουμε να μας περιγράψει τις εμπειρίες της εκεί. Η πρόταση για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, μια που ο κύριος Σοντή έλεγε ότι δεν είναι απαραίτητα ανεξάρτητο, το είπε πριν, εμείς θεωρούμε και εμείς ότι είναι εγγύηση. Συνάδελφε, Ζεατό, σας ευχαριστώ που ε, τονίζετε ότι δεν είναι τρελή η Γερμανία. Είναι πολύ σημαντική η διαπίστωση αυτή, τη συμμερίζομαι. Ωστόσο, ε, θα ήταν κατάχρηση της θέσης μου ως Προέδρου αν ε, έλεγα ποιος αποφασίζει σωστά σε ποιες περιπτώσεις. Ας ελπίσουμε λοιπόν να ε, λειτουργήσει καλά η εσωτερική αγορά. Ε, πριν κλείσουμε το θέμα αυτό, βρίσκεται κανείς εδώ από το Συμβούλιο. Ξέρω ότι στο Συμβούλιο ομάδα εργασίας έχει προσπαθήσει να καταλήξει σε συμβιβασμό στην αρμόδια ομάδα εργασίας. Μήπως θα μπορούσε η Κομισιόν να μας ενημερώσει, μήπως μπορεί να μας πει τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ίσως γνωρίζετε, το Συμβούλιο κάποια στιγμή δυσκολεύτηκε να καταλήξει συμφωνία ανάμεσα στα 25 κράτη-μέλη από τη μία και τα δύο από την άλλη. Η ε, ασυμφωνία αυτή αφορούσε το κομμάτι της σχάσης ε, στο ερευνητικό πρόγραμμα, όχι της ε, σύνδεξης. Ο πρόεδρος της ομάδας υψηλού επίπεδου μαζί με την επόμενη Προεδρία και την Κομισιόν προσπάθησε να καταλήξει σε συμβιβασμό. Μπορώ να σας ενημερώσω ότι χθες επιτεύχθη συμφωνία και ελπίζουμε ότι η Προεδρία θα σας στείλει το κείμενο της, του συμβιβασμού. Με λίγα λόγια, η συμφωνία επιτεύχθη με την επικέντρωση των εθνικών προγραμμάτων περισσότερο στα θέματα ασφαλείας που συνδέονται με όλα τα συστήματα, με τα συστήματα όλων των διαφορετικών καυσίμων. Ε, αυτή η συμφωνία στάλει στην ε, ομάδα εργασίας για την έρευνα τη Δευτέρα. Η Προεδρία ελπίζει, όπως μας είπαν, ότι το πακέτο αυτό θα μπορέσει να σταλεί στην Κορεπέρ στις 22 του μήνα και να υιοθετηθεί την εβδομάδα μετά. Με λίγα λόγια, έχει βρεθεί λύση στο αδιέξοδο με συμβιβασμό. Πιστεύω λοιπόν ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει σύντομα να λάβει σχετική απόφαση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο συνάδελφος Ζιατό και κατόπιν ο κύριος Πρεζίνα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να μας πει αν η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης συμφωνία για τα ποσά. Και έπειτα έχει ληφθεί υπόψη η καταστροφή της Φουκουσίμα. Και ο κύριος Οντί έχει μια ερώτηση ακόμα, παρακαλώ. Ε, Μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, έχει υπάρξει μια επιτάχυνση στο χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου. Εμείς έχουμε την εξασφάλιση ότι το Συμβούλιο θα λάβει γνώση της γνωμοδότησης του Κοινοβουλίου. Γιατί αν ε, δεν μας λάβει υπόψη δεν αξίζει τον κόπο να φτιάχνουμε γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ κύριο Στρόμαγερ. Πρώτη ερώτηση φυσικά. Η συζήτηση στο Συμβούλιο ήταν ε, οι συνέπειες της καταστροφής της Φουκουσίμα, όπως ε, αναφέρθηκε και σας το έχουμε αναφέρει και πριν από λίγες μέρες η συζήτηση εστίασε στο περιεχόμενο και όχι στο προπολογισμό. Σε σχέση με την ερώτηση του κύριου Ντί, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του Συμβουλίου βεβαίως, αλλά Θα το εκτιμούσαμε αν είχαμε την γνώμη της, ε, τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου γρήγορα, ώστε το Συμβούλιο να μπορέσει να το λάβει υπόψη. Μάλιστα. Ο κύριος Συνεμπρεζίνα. Ευχαριστώ όλους όσους πήρατε το λόγο. Από την παρέμβαση του κυρίου Μαντουρέλ την παρέμβαση και την παρέμβαση της σκιώδους ηγήτριας της κυρίας Έρτσοκ προκύπτει το γεγονός ότι όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ είμαι ευτυχής που σας έχω ως ηγήτρια γιατί είστε και μέρος της Επιτροπής ε, προϋπολογισμού, όπου έγινε πολύς λόγος για αυτό το θέμα. Εμείς περισσότερο ασχολούμαστε με το περιεχόμενο, την αξία, την ουσία αυτής της ε, νομοθετικής πρότασης τώρα. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις άλλων συναδέλφων, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Ρούμπικ ότι τα στάνταρ στον τομέα της κατάρτισης και της παιδείας για θέματα που σχετίζονται με την ε, πυρηνική ενέργεια είναι ελλειπής και ε, συμφωνώ και με τους αδέλφους ότι θα έπρεπε να διοργανώσουμε μία ακρόαση Έχουμε το κοινό και ερευνητικό κέντρο, όπως είπε ο συνάδελφος Ζαντό, δεν είναι απόλυτα ανεξάρτητο, αλλά είναι ένας αξιόπιστος οργανισμός, έχει δουλέψει με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά την ακτινοβολία, τον αριθμό των θυμάτων και ούτω καθεξής. Επίσης ήταν παράξενο το γεγονός που στην Ολομέλεια ακριβώς σε αυτή την περίοδο υπήρχε η συζήτηση για τα τεστ αντοχής και δόθηκαν πληροφορίες οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα και όσον αφορά τον κύριο Ποσινόφσκι Εκείνο χρησιμοποίησε το γεγονός Σλαβή για να προωθήσει την έρευνα και τόνισε το γεγονός ότι θετικά χρησιμοποιήθηκαν όλα αυτά. Εγώ στο πλαίσιο των παρατηρήσεών μου για την καταστροφή της Φουκουσίμα θα ήθελα να πω ότι προτείνω ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ ευέλικτο και οι προβλέψεις ε, της είναι επίσης ευέλικτες. Οπότε το θέμα της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας ε, των πυρνικών αποβλήτων, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτή την έρευνα. Επίσης έγινε λόγος για τη σημασία της έρευνας όσον αφορά τη σταδιακή ε, μείωση της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας στη Γερμανία. Ε, εντάξει, η Γαλλία είπε ότι θα συνεχίσει να δίνει την ενέργειά της στη Γερμανία. Δηλαδή, εμείς έχουμε όμως ένα άλλο πρόβλημα, γιατί ε, στις ε, περιοχές όπου υπάρχει εξαιρετική ολική ενέργεια είναι στη Βόρεια Γερμανία. Όμως οι ζώνες κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή η πιο βιομηχανοποιημένη δηλαδή περιοχή, είναι η Νότια Γερμανία. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Η ροή ανάμεσα στη βορρά και στο νότο δεν είναι ομαλή λόγω έλλειψη υποδομών και κάποιες φορές καθώς περνά μέσω της Τσεχίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας η ροή της ηλεκτρικής ενέργειας ε, είχαμε προβλήματα. Κάνω λοιπόν έκκληση στην Γερμανία γιατί είναι λογική η χώρα, λογική Γερμανία, ώστε να κάνουν μια σύνδεση ανάμεσα στο βορρά και το νότο της Γερμανίας. Αλλά εντάξει δεν είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Τώρα, ο συνάδελφος Ζαντό θύμισε πόσο σημαντική είναι η κατάρτιση. Μα όμως αν δεν υπάρχει ποιοτική έρευνα δεν είναι δυνατή η κατάρτιση. Αυτό λοιπόν που δεν κατάλαβα είναι το θέμα που σχετίζεται με την πυρνική έρευνα και τις ιατρικές πτυχές. Εγώ και πιστεύω και ότι και οι ειδικοί δεν μπορούν να φανταστούν ε, πολλαπλές μεθόδους ε, θεραπευτικές χωρίς τη χρήση των ε, πορισμάτων της πυρηνικής ιατρικής έρευνας. Ο συνάλφος Ενέν τώρα υπογράμμισε τις εγγυήσει που, απαιτεί, που απαιτούν οι πληθυσμοί μας όσον αφορά την ασφάλεια. Εγώ θεωρώ ότι ο καλύτερος τρόπος για να εγγυηθούμε ε, αυτά τα στοιχεία είναι οι ρυθμιστές σε εθνικό επίπεδο. Και όσον αφορά την παρέμβαση του κυρίου Ρέμεκ, Συμφωνώ εδώ με τον συνάδελφο Τζιτσέστερ. θα ήταν σημαντικό να προσθέσουμε και άλλους. Στην κεντρική Ευρώπη εμείς καταφέρνουμε να χειριστούμε την παροχή προς την Γερμανία. Και όσον αφορά τις παρεμβάσεις των υπολείπων συναδέλφων, σας ευχαριστώ όλους. Ε, είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι επιτεύχθη μια συμφωνία, ή πιθανότατα από ό,τι φέρετε θα επιτευχθεί η συμφωνία και στο Συμβούλιο. Είμαι βέβαιος ότι και εμείς μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές θα, μπορέσουμε να φτάσουμε σε συνένεση για αυτή την έκθεση και ότι όλα αυτά θα ωφελήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πυρηνική έρευνα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρεζίνα και σημειώνω πρώτον... Α, η Αγγέλη Κανίπλε θέλει πάλι το λόγο, παρακαλώ. Ζήτω συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που διακόπτω. Ε, αλλά ήθελα να αναφερθώ στην έξοδο της Γερμανίας από την πυρηνική ενέργεια που είναι και αυτό ένα θέμα. Ε, ο κύριος Επρεσίν αναφέρθηκε στις δυσκολίες για το τσεχικό δίκτυο. Νομίζω ότι και εσείς έχετε ζητήσει από τον Επίτροπο Oettinger να κάνει ε, μία μελέτη σχετικά με την διαμόρφωση των τιμών τις δυνατότητες του δικτύου. Ήθελα να συμφωνήσω με αυτό και να ρωτήσω εάν ε, η Επιτροπή μας ε, μπορεί να το αναθέσει αυτό σε κάποιον. Ε, έχω συζητήσει και με τον συνάδελφο Ρίπη για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε πληροφορίες και από ε, τον οικονομικό χώρο και θα ήμουν ευγνώμων να μπορείτε να το κάνετε αυτό. Ε, ναι, ίσως θα μπορούσα να το συμπεριλάβω και αυτό στην ε, σύνοψή μου. Πρώτον, λοιπόν, παρακαλούμε την Γραμματεία να εξετάσει το χρονοδιάγραμμα υπό το φως των νέων εξελίξεων στο Συμβούλιο. Δεύτερον, θα παρακαλέσω την Γραμματεία Ε, να μας βρει το αποτέλεσμα της χθεσινής ε, συζήτησης στο Συμβούλιο, διότι αυτό θα μας βοηθήσει να λάβουμε τις αποφάσεις μας ε, πιο γρήγορα. Αν το Συμβούλιο ήδη έχει αποφασίσει, δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να, συζητήσουμε, να συζητάμε κάποια πράγματα. Επίσης, διαπιστώνω ότι ομόφωνα συμφωνούμε στο θέμα της Φουκουσίμα να καλέσουμε κάποιον εμπειρογνώμονα, άσχετα από το τι θα κάνουμε μακροπρόθεσμα για το θέμα αυτό. Θα θέλαμε πολύ να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Φυσικά θα μας απασχολήσει και στο μέλλον το θέμα, αλλά πρώτα να έχουμε μια σύντομη παρουσίαση. Και τρίτον, ευχαριστούμε την ε, Αγγέλη Νίπλερ και τον κύριο Πρεζίνα. Έχω στείλει επιστολή προς τον ε, κύριο Έτιγκερ Πιστεύω ότι θα πρέπει όσο γίνεται πιο σύντομα να ζητήσουμε από την Κομισιόν να μας παρουσιάσει εκείνη τα δικά της αποτελέσματα. Να δούμε ποιες ε, είναι οι συνέπειες ή ποιες μπορεί να είναι. Και ενδεχομένως με τους συντονιστές να συζητήσουμε αν θέλουμε να αναθέσουμε και μελέτη για το θέμα αυτό. Ε, και το θέμα εδώ δεν είναι αν είναι κανεί υπέρ κατά της Γερμανίας. Ε, το θέμα είναι ποιε είναι οι συνέπειες μιας απόφασης σε ένα κράτο μέλος για έξοδο από την πυρηνική ενέργεια και η ενεργειακή πολιτική γίνεται όλο και πιο ευρωπαϊκή και αυτό λοιπόν έχει συνέπειες. Έχουμε συζητήσει και το stress test. Πόσο δύσκολο ήταν να καταλήξουμε τότε σε απόφαση. Δεν καταφέραμε στην Ολομέλεια να υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας. Ε, αυτό ήταν κρίμα. Ε, ε, δεν θα πρέπει να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιες συνέπειες στο μέλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Περνάμε στο επόμενο θέμα της για το πετρέλαιο και φυσικό αέριο ε, δεν ε, θα γίνουν ε, αυτές. Θα πάμε στο θέμα του Γκαλιλαίου. Υπήρξαν συζητήσεις. Από ό,τι γνωρίζουμε βρίσκεται σε καλό δρόμο το θέμα αυτό. Η συγητής έχει πρώτο το λόγο, ο κύριος Γκλάντε. Είχαμε ε, στις 31 Μαΐου τον ε, άτυπο τριμερή διάλογο ε, ήταν ο, ο τρίτος τριμερής διάλογος και μετά από αυτόν τον τρίτο, μέχρι τον τρίτο τριμερή διάλογο είχαμε καταλήξει σε κάποιες συμφωνίες ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Να σας αναφέρω κάποια σημεία κλειδιά όπως είναι η προστασία των δεδομένων. Το Κοινοβούλιο Ε, ζήτησε να γίνει αναθεώρηση γύρω στο 2016. Κατόπιν έχουμε τις ε, διεθνείς ε, συμφωνίες που έχουν ενσωματωθεί που έχουν να κάνουν και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το θέμα της χρηματοδότησης συζητήθηκε έντονα. Το σύστημα Αγκαλιλαίο θα πρέπει να το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο σύστημα, το GPS. Ε, το σήμα θα είναι δωρεάν, ε, αλλά θα πρέπει να ε, εξετάσουμε την συνεισφορά των κρατών χρηστών στο στο, στις, στις δαπάνες, στο κόστος του συστήματος αυτού. Επίσης, ε, όσον αφορά την ασφάλεια του συστήματος, ε, προτείναμε η Κομισιόν να επιβάλλει κυρώσεις ε, όταν δεν θα γίνεται σωστή η χρήση του συστήματος. Το Συμβούλιο δεν το δέχτηκε αυτό. Έχει υιοθετήσει όμως κυρώσεις μέσω των κρατών μελών. Το άρθρο 4, προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων και αυτό ήταν δύσκολο σημείο το Συμβούλιο ε, δέχτηκε την προστασία των δεδομένων αυτών. Αυτή ήταν η κατάσταση κατά τον τελευταίο τριμερή διάλογο. Και ο Πρόεδρος, ο κύριος Ρόιλ και εγώ καταφέραμε να συμφωνήσουμε σχετικά με τα τελευταία σημεία. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Ε, συζητήσαμε τις κατεξουδότηση πράξης ε, που είναι πάντα ένα αγαπημένο θέμα. Υπήρξε έντονη συζήτηση σχετικά με το άρθρο 8. Το Συμβούλιο έχει αποδυναμώσει την αρχική πρόταση για να αποφύγει της κατεξουσιδότηση πράξης. Ε, και το Κοινοβούλιο θα επηρεαστεί από αυτό. Υπήρξε εδώ σημαντική διαφωνία. Η Κομισιόν είχε προσθέσει ένα μεγάλο παράρτημα των θεμάτων που θα ε, άλλαζε με κατεξουδότηση πράξης. Ε, το Συμβούλιο να τον κατάλογο αυτό. Τελικά ε, καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό. Το Κοινοβούλιο δέχεται το συντομευμένο αυτό παράρτημα. Ωστόσο, η τροποποίηση μέσω πράξεων κατοξιδότηση μπορεί να γίνει. Επίσης υπήρξε μια δήλωση του Συμβουλίου, υπήρξε μια δήλωση την οποία ε, συζητήσαμε πολύ έντονα χθες. Το θέμα ήταν σε τι βαθμό τα κράτη-μέλη ε, θα υποχρεώνονται από αυτά που λέει η Κομισιόν. Τελικά καταλήξαμε σε έναν συμβιβασμό. Γενικά πάντως ε, μετά την εχθεσινή συζήτηση καταλήξαμε σε συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν και έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή την νομοθεσία κατά την πρώτη ανάγνωση. Ωστόσο, η ψηφοφορία ε, στην Ολομέλεια μάλλον θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Πάντως η Ουγγρική Προεδρία κατάφερε να πετύχει το συμβασμό αυτόν. Ευχαριστούμε την Προεδρία. Σίγουρα δεν θα ήταν πολύ εύκολο ο συμβασμό αυτόν. Ε, θα υπήρχαν σίγουρα κρατημέλη, δεν λέω ονόματα, που θα είχαν φέρει σημαντικέ αντιρρήσει. Πάντω τα καταφέραμε. Θα σας πω αυτό που είπα και στον τριμερή διάλογο. Ε, αυτό που, στο οποίο θα επιμείνουμε δεν είναι η συμφωνία στην ε, πρώτη ανάγνωση, ε, αλλά αν μπορούμε να την πετύχουμε φυσικά αυτό είναι καλό. Πάντως δεν θα πρέπει να γίνει αυτός ο κανόνας, ε, θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κλάντε και τους ε, συνεργάτες του. Ευχαριστώ και τους συναδέρφους για την ε, καλή συνεργασία. Άλλωστε φαίνεται και το αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε, αλλά αυτό είναι καθαρά τεχνικό θέμα, θέμα διαδικασίας. Στις 30 Ιουλίου θα ψηφίσουμε τελικά. Ήταν καλό το αποτέλεσμα και η Ουγγρική Προεδρία σίγουρα έχει συμβάλει. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε μία μελέτη για ένα θέμα που μας απασχόλησε και χθες. Την στρατηγική της ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο, στη Νότια Μεσόγειο. Θα παρακαλούσα τους ομιλητές ε, να έρθουν εδώ. Λοιπόν, έχουμε εδώ το θέμα ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεσογειακό Νότο. Έχουμε αναθέσει η εκπόνηση μελέτης τον Ιούνιο του 2010 ε, το αποφασίσαμε και τον ε, Μάρτιο του 2011 ε, παρουσιάστηκε το αποτέλεσμα. Θα παρουσιαστεί λοιπόν η μελέτη από δύο εμπειρογνώμονες τους οποίους καλωσορίζω θερμά, τον κύριο Μπερνάρντιο Αρμέλ, ελπίζω να προφέρω σωστά τα ονόματα, και τον Henri Μπουσόν. Ελπίζω να τα είπα σωστά. Α, ευχαριστώ πολύ, μου λέτε ότι τα λέω καλά. Και... Τώρα ενδιαφερόμαστε όλοι για τα πορίσματά σας. Σειρά σα. Euh, euh, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Bernard Duhamel. Αν μου το επιτρέπετε θα μιλήσω στα γαλλικά, τη μητρική μου γλώσσα. Θα ξαναεκκρινίσουμε λοιπόν αυτή την παρουσίαση με τον συνάδελφο Henri Bosson και θα σας παρουσιάσουμε και αυτές τις διαφάνειες. Για τη Μεσόγειο λοιπόν, εδώ ο χάρτης αυτό σας δείχνει την ε, γεωπολιτική σημασία του συνόλου. Εκτείνεται σε τρεις υπήρους. Βρέχει τρεις υπήρους η Μεσογειακή Λεκάνη. Εντάξει, εδώ έχετε μια εικόνα της μεσογειακής ζώνης. Αυτό στόχο έχει να σας δείξει ποιες είναι οι χώρες, οι περιοχές στις οποίες έχουμε για τις οποίες έχουμε εργαστεί. Η μελέτη μας αφορά λοιπόν τη Μεσογειακή Λεκάνη στο σύνολό της, πράγμα που συμπεριλαμβάνει χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στη βόρεια όχθη της Μεσογείου και τις χώρες του Νότου και της Ανατολικής Μεσογείου Κατά βάση ασχοληθήκαμε με τις μεσογειακές χώρες, είναι 7, αλλά προσθέσαμε και την Πορτογαλία, η οποία επειδή βρίσκεται στην Ιβηρική Χερσόνησο θεωρείται παραδοσιακά μεσογειακή χώρα. Έχουμε λοιπόν την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Ελλάδα, συν Κύπρος και Μάλτα. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η Μάλτα και η Κύπρος δεν έχουν φυσικό αέριο. Η Μάλτα μάλλον δεν πρόκειται και να γίνει ποτέ χώρα που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο λόγω του κόστους. Ε, αντίθετα για την Κύπρο υπάρχει ένα σοβαρό πρόγραμμα κατασκευής ενός ε, ε, εργοστασίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και έπειτα νότιος έχουμε το Μαρόκο μέχρι και την Τουρκία με το Μαγκρέμπ, Μαρόκο, Αλγερία, την Ισία, τη Λιβύη που δεν ανήκει τουλάχιστον ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση και το σύνολο Μασρέκ, ΡΕΚ, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, η Ορδανία που ούτε και αυτή αυστηρά βρέχεται από τη Μεσόγειο αλλά που θεωρείται ως τμήμα των μεσογειακών χωρών και του Μασρέκ είναι μάλιστα μία από τις χώρες που εντάσσονται στο Master Plan Φυσικού Αερίου το Ευρωασιατικό και μαζί έχουμε την Τουρκία και το Ισραήλ. Και ε, τούτο ο χάρτη είναι σίγουρα νέο, είναι, είναι νέο για κάποιου από εσά. Δείχνει το βυθό τη Μεσογείου θάλασσα. Γιατί, Γιατί πρέπει κανεί να διασχίσει τη Μεσόγειο θάλασσα με τους αγωγούς φυσικού αερίου αλλά και με προγράμματα που μπορεί να φτιαχτούν και να αφορούν την μεταφορά ρεύματο. Ε, και όπως βλέπουμε, και δεν το γνωρίζουμε αρκετά, η Μεσόγειο στα ορισμένα της κομμάτια είναι εξαιρετικά βαθιά. Προς Ανατολάς, ε, η βυθή που είναι με σκούρο γαλάζιο είναι βάθος λιγότερο από 3.000 μέτρα. Μέχρι 5.000 μέτρα φτα... βάθος φτάνει η Μεσόγειος θάλασσα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλα φυσικά προβλήματα τα οποία δεν είναι διόλα μελιτέα. Τώρα, για να τελειώσουμε αυτήν την εισαγωγή όσον αφορά τις συγκρίσεις που μπορούμε να κάνουμε ανάμεσα στο βορρά και στο νότο της Μεσογείου Θα λέγαμε ότι από δημογραφικής άποψης αυτή τη στιγμή πρόκειται για πληθυσμούς συγκρίσιμους, 200 εκατομμύρια κάτοικοι από την κάθε όχθη. Αντιθέτως, ο νότος της ε, Μεσογείου ωστόσο αυξάνεται τέσσερις φορές πιο γρήγορα, πληθυσμιακά αυξάνεται τέσσερις φορές πιο γρήγορα από ότι ο βορράς της Μεσογείου. Και όσον αφορά τις διαφορές στην κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση κατά κεφαλήν ηλεκτρικής ενέργειας στον Βορρά είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από ό,τι στον Νότο. Έχετε τα νούμερα ε, με διαφέρουν από χώρα σε χώρα, κυρίως στην ε, νότια όχθη. Μόνο μία χώρα φαίνεται να είναι ισότιμη με τις βόρειες χώρες, είναι το Ισραήλ. Οι υπόλοιποι Στο Μαρόκο, για παράδειγμα, έχουμε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πραγματικά πολύ χαμηλή. 600 κιλοβατόρες κατά κεφαλήν. Oui, alors juste euh, quelques chiffres, sans vous bien sûr avec des chiffres. Κάποια αριθμητικά στοιχεία, δεν θέλω να σας κουράσω βέβαια με αριθμούς, αλλά κάποια στοιχεία πρέπει να σας δώσω. Για το φυσικό αέριο να σας πω κάποια στοιχεία γιατί ο Μπερνάρ ο ειδικό για την ε, ηλεκτρική ενέργεια, την αποτελεσματικότητα, την απόδοση του ηλεκτρισμού κτλ. Ενώ εγώ περισσότερο για το φυσικό αέριο. Λοιπόν, για το φυσικό αέριο θα πρέπει να δούμε ότι η κατανάλωση ε, φυσικού αερίου, και εδώ σας δίνω στοιχεία του 2009, τη στιγμή που συντάξαμε την έκθεση δεν είχαμε ακόμα τα στοιχεία για το 2010, πάντως στις ε, μεσογειακές χώρες στην Ευρωπαϊκή Μεσόγειο το φυσικό αέριο ανέρχεται στο ίμιση των εισαγωγών του συνόλου του εισαγωγών φυσικού αερίου ολόκληρη της Ευρώπης. Γιατί? Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να πούμε ότι αντίθετα με τα όσα συμβαίνουν για άλλες πρωτεσίλες, τα αποθέματα και παραγωγή είναι στο βορρά και όχι στο νότο. Στις χώρες λοιπόν τις Μεσόγειακές μόνο μία χώρα είναι σημαντικός παραγωγός φυσικού αερίου, η Ιταλία. Αλλά διαφορετικά στις υπόλοιπες νότιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε τους όγκους φυσικού αερίου που έχουμε στο βορρά της Ευρώπης, ειδικά στην Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία και στην Πολωνία συν τις ε, χώρες ε, της Βαλτικής που είναι σημαντικός ε, εισαγωγές. Η εξάρτηση λοιπόν των νότιων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από... είναι της τάξης του 95%. Σημαίνει αυτό δηλαδή ότι το μεγαλύτερο τμήμα του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στις νότιες χώρες εισάγεται. Η παραγωγή δε φυσικού αερίου μειώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάποιες χώρες έχει σταματήσει τελείως, όπως στην Ισπανία και στη Γαλλία. Μόνο έχει μείνει η Ιταλία στην Νότια Ευρώπη. Μπορούμε να θεωρήσουμε δηλαδή ότι σε ορισμένες χώρες, μάλλον σε ορισμένα χρόνια, το φυσικό αέριο που θα καταναλώνεται στις νότιες χώρες θα είναι απόλυτα εισαγόμενο. Εδώ έχετε το σχέδιο τώρα της παρουσίασής μας. Έχουμε λοιπόν τις ευρωπαϊκέ πολιτικές που θα σας παρουσιάσουμε καταρχήν, την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και διάφορες συστάσεις που προκύπτουν από αυτή τη μελέτη. Ας περάσουμε λοιπόν στις πολιτικές της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Πρόκειται για βασικέ γραμμέ, τι οποίε γνωρίζετε κι εσεί και ίσω και καλύτερα από εμά. Αυτό που ήθελα εγώ να ε, αναφέρω σε αυτή την πρώτη διαφάνεια είναι ένα από τα πρόσφατα δημιουργήματα, μία από τι οδηγίε που είναι η δημιουργία των ENCHO E ε και ENCHO G, που είναι τα ευρωπαϊκά ε, δίκτυα για τους ε, φορείς ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Αυτά δημιουργήθηκαν λοιπόν ε, για να έχουμε σχέδια υποδομών, να φτιάξουμε σχέδια υποδομών έτσι ώστε να υπάρχει σχεδιασμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο φτιάξαμε και τα δεκαετή προγράμματα για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Κάθε δύο χρόνια ανανεώνονται αναθεωρούνται. Εν γέννη δηλαδή είναι στο τέλος των ε, ζυγών χρονιών, δηλαδή το πρώτο έγινε, έγινε η πρώτη αναθεώρηση το 2008, το δεύτερο το 2010. Οι, στρα, οι προτεραιότητες Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό γιατί η στρατηγική του Νοεμβρίου 2010 είναι η ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ευρωπαϊκής αγοράς και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να υπάρξει ολοκλήρωση όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ολοκλήρωση των αγορών ενέργειας και με τον Νότο. Περιφερειακή δηλαδή ολοκλήρωση των αγορών ε, ενέργειας του Νότου. Είδαμε ότι AMGNP είναι μια διοίκηση, αλλά να υπάρχει πιο προωθημένη συγχώνευση των αγορών ε, της Ευρώπης με τις αγορές της ε, Νότιας Μεσογείου. Ενδιαφέροντος αυτός ο χάρτης. Διότι από τη μια πλευρά τονίζει και αξιοποιεί κάτι που δεν είχε γίνει παλιότερα, τους ενεργειακούς διαδρόμους, τους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας δηλαδή, από τη μια πλευρά στο εσωτερικό της Ευρώπης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ενιαία αγορά και να μπορέσουν και χώρες που δεν ε, είναι ευνοημένες από άποψη πρώτων υλών και ενέργειας να υποφεληθούν από την ενέργεια σε άλλες χώρες, από τους πόρους σε άλλες γειτονικέ χώρες και έπειτα έχετε και τους ενεργειακούς διαδρόμους ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την όχθια, όχθη της Μεσογείου. Έχουμε δηλαδή τον νότιο διάδρομο έτσι όπως αποκαλείται που θα πρέπει να επιτρέψει στους πόρους της Μέσης Ανατολής να φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ανατολή και από τον Νότο. Euh, euh, και έχουμε και τον Ανατολικό Διάδρομο για τις ανταλλαγές ηλεκτρισμού. Από αυτές τις ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να επιμείνουμε στην οδηγία για την ανανεώσιμη ενέργεια, την οποία σίγουρα γνωρίζετε. Αυτή ορίζει στόχους 20% ε, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για το 2020. Θα πρέπει επίσης ε, όσον αφορά την σχέση βορανότου να επιμείνουμε στο άρθρο 9, το οποίο έχει πολύ συζητηθεί εξάλλου, που προβλέπει ότι κοινά προγράμματα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις τρίτες χώρες πράγμα που θα επέτρεπε να υπάρξει παροχή ενός σημαντικού όγκου ανανεώσιμης ενέργειας από τις ε, χώρες του Νότου. Πράγμα το οποίο υποδεικνύει ότι οι ευρωπαϊκοί στόχοι μπορούν ε, να διευκολύνουν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις νότιες χώρες, δηλαδή Μαρόκο, Συρία, ας πούμε, περνώντας από την Αίγυπτο. Όσον αφορά τώρα τον ηλεκτρισμό. Διάδρομος για την εξαγωγή τα βλέπετε εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια. Είναι οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, Αλγερία, Μαρόκο, Τινησία, Μαγκρέμπ δηλαδή, Προ την Ισπανία που υπάρχει ήδη η σύνδεση και προς την Ιταλία που είναι ένα σχέδιο. Γιατί πρόκειται για μια σύνδεση ανάμεσα στην Τινησία και την Ιταλία κυρίως και έπειτα υπάρχουν και άλλες δυνατότητε σύνδεση. Και θα δούμε στη συνέχεια τι δυσκολεύει την πραγματοποίησή τους. Ανάμεσα δηλαδή στις χώρες ανατολικά τη Μεσογείου και τα Βαλκάνια. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των Βαλκανίων. Το σύνολο τώρα των διασυνδέσεων στην Μεσόγειο έχουν να κάνουν με το μέντερινγκ. Βλέπουμε εδώ ποιες είναι οι συνδέσεις που υπάρχουν εδώ πέρα. Είμαστε από το 2008 ε, και είναι σε γίγαβατ. αν δείτε στο Νότο, οι συνδέσεις αυτές είναι πολύ πιο λίγες και υπάρχει και κατακαιρματισμός των συνδέσεων αυτών. Κατακαιρματισμός με τρεις πόλους. Τον ε, πόλο της Βόρειας Αφρικής, των χωρών Μαγκρέπ, που κόβεται από τη σύνδεση την Ισία Λιβύη, εκεί δηλαδή δεν γίνεται καλά. Υπάρχει ένας άλλος πόλος με κέντρο την Αίγυπτο και υπάρχει και ο πόλος Τουρκία που ήδη ενσωματώνεται πολύ περισσότερο στο ευρωπαϊκό σύνολο. Και γι' αυτό είναι αποκομμένος από ε, την ε, σύνδεση με την Αίγυπτο και με τη Συρία κλπ. Έρχομαι τώρα στον πόλο των χωρών Μαγκρέμπ. Να, πώς έχουν οι συνδέσεις, το βλέπετε εδώ στη διαφάνεια αυτή. Είναι οι τρεις χώρες και η Ισπανία. Υπάρχει μια διπλή σύνδεση μεταφοράς ηλεκτρισμού από την Ισπανία στο Μαρόκο. Το Μαρόκο εισάγει ηλεκτρισμό. Και έπειτα υπάρχουν και συναλλαγές με διασυνδέσεις ανάμεσα στο Μαρόκο, την Αλγερία και την Τινησία. Και βλέπουμε εδώ ότι η Δινησία με την Λιβύη υπάρχει, αλλά είναι πολύ αδύναμη. Και λειτουργεί πάρα πολύ άσχημα. Έρχομαι στον ε, τουρκικό τώρα ενεργειακό πόλο. Εδώ υπάρχουν τρεις συνδέσεις με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία όπου η σύνδεση Ελλάδα-Βουλγαρία-Τουρκία, η ενεργειακή κοινότητα δηλαδή αυτή μεταξύ Βαλκανίων και Τουρκίας, γίνεται ο συγχρονισμός και θα ολοκληρωθεί το 2012. Ο όρος, η προπόθεση για να γίνει, είναι να διακοπεί ο συγχρονισμός με τη Συρία. Πράγμα που σημαίνει ότι το 2015, ίσως και αργότερα, θα έχουμε τη σύνδεση Τουρκίας με την υπόλοιπη Νότια Μεσόγειο. Εδώ βλέπουμε ένα σχήμα που δείχνει τον πόλο της Αιγύπτου, που έχει στρατηγική θέση. Η, Αιγύ... η Αίγυπτος με 80-85 εκατομμύρια κατοίκους, καταλαβαίνετε ότι έχει μεγάλο βάρος. Και οι ενεργειακές της ανάγκες αυξάνονται πολύ. Το ενεργειακό της σύστημα είναι πλήρες και οι ανάγκες της, όπως είπαμε, είναι μεγάλες. Συνεπώς, η Αίγυπτος θα πρέπει και αυτή να τροφοδοτείται. Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον ε, προμήθειες μέσω του Νείλου με έργα που γίνονται στην Αιθιοπία. Αλλά υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης Αιγύπτου-Αιθιοπίας. Υπάρχουν και ε, δυνατότητες από τις χώρες του κόλπου. Αλλά και εδώ υπάρχουν προβλήματα, επειδή ίσως δεν φτάνουν όλα αυτά. Πρέπει να ξέρουμε ότι η δημογραφική εξέλιξη στην Αίγυπτο σημαίνει ότι αυξάνονται πάρα πολύ, αυξάνεται πάρα πολύ ο πληθυσμός στη χώρα αυτή. Οι ενεργειακές ανάγκες λοιπόν θα πολλαπλασιαστούν. Και αυτό πρέπει να λυθεί γιατί η δημογραφική εξέλιξη σημαίνει ε, περισσότερος κόσμος στις πόλεις, πράγμα που σημαίνει περισσότερο νερό στις πόλεις και περισσότερο νερό στις πόλεις σημαίνει μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση. Το 2005 θα έχουν φτάσει 150 εκατομμύρια Αιγύπτιοι. Οι τρεις χώρες λοιπόν Μαγκρέπ είναι αυτές που έχουν ε, τις πιο μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης εν ώψη του 2020 εξαιτίας της σύνδεσης με την Ισπανία πάνω απ' όλα και εξαιτίας και συνδέσεων που θα γίνουν με την Ιταλία όπου έχουμε το ΕΛΜΕΔ, την Ισία Ιταλία, είναι το πιο προχωρημένο πρόγραμμα, το οποίο γύρω στο 2016 προβλέπεται να ολοκληρωθεί. Είναι ένα πρόγραμμα, υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα μάλλον, Αλγερία Ιταλία μέσω της Σαρδινίας για αργότερα. Είναι σχέδιο ακόμα. και περιμένουμε να υπάρξει και ενίσχυση των ε, διασυνδέσεων Μαρόκο, Αλγερία, την των τριών αυτών αγορών. Υπάρχει ένα σχέδιο ολοκλήρωση ε, της ενεργειακής αγοράς ε, στις χώρες Μαγκρέπ. Είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δήλωση για να ενισχυθεί η συνεργασία των τριών αυτών χωρών στον τομέα της ενέργειας. Οι τρεις Υπουργοί Ενέργειας συναντήθηκαν στο Αλγέρι την παρουσία του Επιτρόπου του Αρμόδιου για την Ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις Βρυξέλλες επίσης τον Οκτώβριο έγινε μία επαφή και τον Απρίλιο ήταν στο Αλγέρι. Τώρα το μεσογειακό σχέδιο για την ηλιακή ενέργεια. Προσπαθούμε να πετύχουμε λύσεις, να βρούμε λύσεις στο ενεργειακό πρόβλημα, επειδή η ζήτηση στις νότιες χώρες, η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται κατά πολύ. Θέλουμε με 20 γίγαβατ να προχωρήσουμε, με μια επιπλέον δηλαδή, ένα επιπλέον δυναμικό 20 γιγαβάτ. Με τα φωτοβολταϊκά, με την ηλιακή ενέργεια, την συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια, θερμική και την αιωλική ενέργεια που υπάρχει άφθονη στις χώρες του Νότου. Τα κύρια κέντρα είναι στο Μαρόκο και την Αίγυπτο. Υπάρχει αιωλική ενέργεια. Υπάρχουν δυνατότητες για αιωλική ενέργεια βέβαια και στην την Ισία, αν και μικρότερες. Ένας άλλος στόχος του σχεδίου αυτού για την Μεσόγειο είναι ότι υπάρχουν εξελίξεις τέτοιες που μας επιτρέπουν περισσότερο τη χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας με συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα. Οπότε εμφανίζονται οι ιδιωτικές επενδύσεις που στηρίζουν αυτό το στόχο. Αναπτύσσεται λοιπόν μια ολοκληρωμένη αγορά ευρωμεσογειακή, μια που ένας από τους στόχους είναι αυτός ο ηλεκτρισμός από την ηλιακή ενέργεια εν μέρη να φτάσει στην Ευρώπη. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να λυθούν τα τεχνικά ζητήματα που τίθενται όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια και έχουν να κάνουν με, διαφορε... με το γεγονός ότι δεν έχουμε πει μονίμου βάσεως την ίδια παραγωγή γιατί τον ήλιο δεν τον έχουμε πάντα εξίσου. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παράγεται όταν έχουμε τον ήλιο. Υπάρχει και η γερμανική πρωτοβουλία, Desert Tech λέγεται, η οποία ξεκίνησε το 2009. Λίγο μετά την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Είναι μια ιδιαίτερα φιλόδοξη πρωτοβουλία αυτή, η οποία προβλέπει την παραγωγή για το 2050 μερικών εκατοντάδων γιγαβάτ με επενδύσεις που αρχικά εκτιμήθηκαν στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η πρωτοβουλία καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι της ε, ερήμου, γιατί βλέπετε ότι στην έρημο κυρίως έχουμε την ηλιακή ενέργεια, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση. Συνοδεύεται όμως και από μια άλλη πρωτοβουλία γιατί πρέπει να μεταφερθεί στη συνέχεια ο ηλεκτρισμός αυτός. Πρέπει να διασχίσει την Μεσόγειο, εφόσον θέλουμε να φτάσει στην Ευρώπη κάποια στιγμή. Και έτσι έχουμε το Μεγκρίν. Είναι το consortium MedGrid. Είναι γαλλική πρωτοβουλία πρόσφατη αυτή. Επισημοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες μόλις. Και έτσι ξεκίνησαν ε, μελέτες σκοπιμότητας για να δούμε κατά πόσο μπορεί να έρθει αυτό το φυσικό κατά κάποιο τρόπο εμπόδιο που είναι η Μεσόγειος, εμπόδιο στη μεταφορά του ηλεκτρισμού. Τα πρώτα αποτελέσματα θα τα έχουμε το 2013. Πρόκειται, όπως σας είπα, για μελέτες σκοπιμότητας. Υπάρχει τώρα και μια άλλη σημαντική πτυχή για την ευρωπαϊκή πολιτική και για την ανάπτυξη της ενεργειακής πολιτικής των χωρών αυτών του Νότου και είναι η πρόθεση της ενεργειακής απόδοσης. Διαπιστώνουμε ότι η ενεργειακή απόδοση ε, προχωράει στις χώρες του Βορρά και στις χώρες του Νότου, αλλά διαπιστώνουμε ότι η πρόοδος στη δεύτερη κατηγορία χωρών δεν είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που διαπιστώνεται στις χώρες του Βορρά. Συνεπώς πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες προσπάθειες, να στηρίξουμε δηλαδή τις χώρες του Νότου με ε, νομοθεσία. Κάτι το οποίο έχουν αρχίσει να κάνουν οι χώρες αυτές, το Μαρόκο, η Αίγυπτος, η Ισία, η Ορδανία, έχουν υιοθετήσει νομοθετικές διατάξεις και το Ισραήλ προς αυτήν την κατεύθυνση. με αυτές τις ενεργειακές εξελίξεις που πάμε. Η βασική ιδέα είναι να φτάσουμε σε ένα σούπερ δίκτυο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Ένα δίκτυο το οποίο θα βασίζεται σε ένα σχέδιο εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορούμε να διασχίζουμε τη θάλασσα μέσω αυτού του δικτύου χωρίς δυσκολίες και χωρίς να ε, καταφεύγουμε πάντα στη λύση Γιβραλτάρ. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν ε, γραμμές υψηλής τάσεως, direct, direct, για μεγάλες αποστάσεις, που θα χρησιμοποιούνται ως άξονες. Το πρόβλημα είναι πάντα πως αυτήν την ενέργεια που όπως είπαμε δεν είναι σταθερής ροής από τις ε, εναλλακτικέ μορφές ενέργειας, είτε πρόκειται για την ηλιακή είτε την αιωλική και όπως είπαμε η αιωλική δεν είναι τόσο σημαντική, αν και υπάρχουν δυνατότητες στο κόλπο του Σουέζ. Μιλάμε κυρίως εδώ για την ηλιακή, που όπως είπαμε δεν έχει συνεχή ροή. Τα δίκτυα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα και πλήρη. Άρα φτάνουμε σε ένα, πώς το πω, σε ένα κρίκο που έχει τη μορφή λίγο πολύ αυτή που βλέπετε σε αυτή την διαφάνεια. Βλέπετε Ιταλία και οι γείτονες χώρες. Η Ιταλία και εισάγει και έστελνε ενέργεια πολύ. Έρχομαι τώρα στο φυσικό αέριο. Για το φυσικό αέριο. Η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Εδώ έχουμε ζητήματα και όσον αφορά την παραγωγή, μάλλον όχι, για το ηλεκτρικό. Έχουμε το πρόβλημα και στην παραγωγή και στις υποδομές, ενώ για το φυσικό αέριο, δε το φυσικό αέριο υπάρχει, τα προβλήματα που καλούμε θα αναλύσουμε είναι τα προβλήματα μεταφοράς και ασφάλειας εφοδιασμού. Θα σας δείξω εδώ έναν ενδιαφέροντα χάρτη γιατί δείχνει τις ζώνες επιρροής ποιοι είναι οι κύριοι εξαγωγής φυσικού αερίου σήμερα προς την Ευρώπη. Βλέπετε το μεγάλο πορτοκαλί κομμάτι δεξιά που είναι η Ρωσία. Το πράσινο δυτικά είναι οι εισαγωγέ από την Αλγερία βασικά. Και μετά βλέπετε το μπλε κομμάτι που είναι η Νορβηγία, κυρίως και βαλτικές χώρες. Η Ρωσία φυσικά έχει τεράστιο όγκο, το βλέπετε. Είναι οι τέσσερις μεγάλοι προμηθευτές ε, φυσικού αερίου προς την Ευρώπη σήμερα. Βέβαια δεν είναι απόλυτα ακριβής ο χάρτης, γιατί, γιατί δείτε την Ιταλία, η Ιταλία δείχνει να προμηθεύεται αποκλειστικά από την Ρωσία φυσικό αέριο, ενώ τώρα προμηθεύεται και από τη Λιβύη και από την Τινησία σε μεγάλο βαθμό. Τώρα πώς ε, έρχεται και πώς μεταφέρεται το φυσικό αέριο με αγωγούς φυσικού αερίου που είναι υποθαλάσσιοι, γιατί πρέπει να διασχίουν την Μεσόγειο. Εδώ βλέπετε κάποια σχέδια και τις ε, συνδέσεις που ήδη υπάρχουν. Υπάρχουν τρεις αγωγοί που συνδέουν την Αλγερία, την Αλγερία και την ε, Λιβύη με την Νότια Ευρώπη επίσης μέσω της Αλγερίας προς την ε, Ισπανία και άλλοι δύο από την Αλγερία πάνε στην Ιταλία μέσω της Σικελίας. Και υπάρχει και ο πράσινος που βλέπετε δεξιά σας, που είναι ο πιο πρόσφατος αγωγός και που φέρνει φυσικό αέριο από τη Λιβύη. Και υπάρχουν και δύο σχέδια, δύο σχέδια τα οποία δεν λειτουργούν ακόμα βέβαια που συνδέουν την Ισπανία με την Αλγερία έχει μπει ο αγωγός αλλά δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Γιατί η αγορά κατέρευσε από το 2009 και οι Ισπανοί δεν βρίσκουν πελάτες για το φυσικό αέριο που θεσάγουν. Και σε πορτοκαλί βλέπετε μέσω ε, Σαρδινίας και Κορσικής συνδέουμε την Αλγερία με την Ιταλία. έχουμε εντοπίσει τρία κύρια προβλήματα. Και τα τρία έχουν να κάνουν με την διασφάλιση του κύριου στόχου, δηλαδή την ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου. Αυτό είναι το light motive. Δηλαδή αν ένα πράγμα πρέπει να συγκρατήσει κανείς από όλη μας τη μελέτη είναι ότι πρέπει έτσι κι αλλιώς να υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί, γιατί το βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο θα εισάγουμε φυσικό αέριο, ιδίω οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, το είδαμε ότι κατά 95% εξαρτώνται από εισαγωγές φυσικού αερίου οι χώρες της Νότιας Ευρώπης. Συνεπώς χρειάζεται διαφοροποίηση των πηγών από όπου προμηθευόμαστε φυσικό αέριο. Και πώς ξεκινάμε με τις τεχνικές και οικονομικές ε, εξελίξεις όσον αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είπαμε, έχει πολλά θετικά το φυσικό αέριο, αλλά από την άλλη μεριά το υγροποιημένο μπορεί να έρθει με πλοία και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τελευταία. Όσον αφορά την προμήθεια, έχουν υπάρξει τεράστιες εξελίξεις και τώρα υπάρχουν κάπου 15 χώρες που προμηθεύουν αέριο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, ενώ την δεκαετία του 80 είχαμε το πολύ 12 με τις τέσσερις μεγάλες που είναι Νορβηγία, κάτω χώρες, Αλγερία και Ρωσία. Ενώ τώρα γίνεται αυτή η διαφοροποίηση. Δεν φτάνει όμως ακόμα. Και δεν φτάνει γιατί οι ανάγκες αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Ακόμα και αν συνεχίσουν να αυξάνονται λιγότερο από ό,τι έχει γίνει ε, τον τελευταίο καιρό εξαιτία και άλλων εναλλακτικών πηγών ενεργειών, αλλά μην ξεχνάμε ότι το φυσικό αέριο χρησιμεύει για την παραγωγή ηλεκτρισμού στην Ευρώπη σε ένα μεγάλο βαθμό. Οπότε, ακόμα και αν η ζήτηση δεν αυξάνεται ακόμα τόσο πολύ όσο αυξήθηκε πρόσφατα, παρόλα αυτά χρειάζεται να βρούμε τρόπους διασφάλισης του εφοδιασμού Ακόμα και αν φτάσουμε μέχρι το Ιράκ, Ιράν, Κασπία, Περσικό κόλπο, όλες αυτές είναι πηγές που κατεξοχήν μπορούν να εξυπηρετούν την Ευρώπη. Να εδώ ένα σχέδιο το οποίο σας δείχνει ποια είναι τα σημερινά σχέδια για να έχουμε φυσικό αέριο από ε, το τμήμα ανατολικά της Μεσογείου. Υπάρχουν δύο βασικά σχέδια. Υπάρχει το Ναμπούκο σε κόκκινο, που σωστά υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που φέρνει φυσικό αέριο είτε από το Αζερμπαϊτζάν, είτε από το Ιράκ, είτε από το Ιράν, εφόσον η πολιτική κατάσταση εκεί είναι τέτοια που να το επιτρέπει. Κεντρική Ευρώπη επίσης και φτάνουμε και στα σύνορα Αυστρίας-Ουγγαρίας. Είναι το πιο παλιό σχέδιο αυτό. Έχει ήδη δύο χρόνια και συμπληρώθηκε από ένα ρωσικό-ιταλικό σχέδιο στο οποίο συμμετέχουν τώρα και οι Γάλλοι, η ΕΝΤΕΦ, που λέει μέσω της ε, Μαύρης Θάλασσας να φτιάξουμε έναν αγωγό από τη Ρωσία προς την Βουλγαρία. Και υπάρχουν και άλλα δύο που είναι Ελλάδα-Ιταλία όπου φέρνουμε δηλαδή στην Ιταλία από το Αζερβαϊτζάν φυσικό αέριο και μετά πάει στην Βόρεια Ευρώπη. Από σχέδια έχουμε πολλά. Και γιατί υπάρχει το Ναμπούκο και το South Stream και μοιράζεται ο κόσμος ανάμεσα στα δύο. Αυτά τα δύο μπορούν να καλύψουν την ενδυνάμει ζήτηση, την αυξανόμενη που αναμένουμε για χρόνια και για δεκαετίες. Είναι ανταγωνιστικά λοιπόν αυτά τα δύο δίκτυα μεταξύ του. Είναι θέμα στρατηγική και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα το δούμε. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, εν Γιατί, Γιατί τον, Ναμπούκο, τον Ναμπούκο που ήταν το πρώτο και που κατά τη γνώμη μου έχει περισσότερο νόημα, φτάνει να διασφαλίσει τον εφοδιασμό για πάρα πολλά χρόνια. Άρα με κάποια συμπληρώματα θα φτάνε. Το πρόβλημα όμω είναι ότι η Ρωσία που εξακολουθεί να είναι ο πιο σημαντικός προμηθευτής φυσικού αερίου για την Ευρώπη, έχει ξεκινήσει το South Stream, το δικό της πρόγραμμα. Και δεν θέλει επιπλέον πηγές ε, για την Ευρώπη. Δεν θα δηλαδή η Ευρώπη να καταφεύγει στο Αζερμπαϊτζάν ή στο Ιράκ. Γι' αυτό λέω ότι είναι ανταγωνιστικά αυτά τα δύο προγράμματα, το Ναμπούκο με το South Stream. Από όσο ξέρω δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία ε, απόφαση, αλλά σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα. Αν θέλουμε πραγματικά ε, διαφοροποίηση, πρέπει η διαφοροποίηση να υπάρχει στην πηγή. Το μόνο σχέδιο το οποίο βελτιώνει τη διαφοροποίηση είναι το Ναμπούκο. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ωραία, λοιπόν. Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι, ωραία, θέλουμε να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την αύξηση των αναγκών στις χώρες προμηθευτές. Κάτι το οποίο προς το παρόν δεν έχει ληφθεί υπόψη από την Ευρώπη. Δηλαδή, για να έχουμε μια τέτοια ανάπτυξη ε, προμήθεια στην ε, Ευρώπη, πρέπει να έχουμε ανάπτυξη της παραγωγής και στις χώρες που μας προμηθεύουν φυσικό αέριο. Οι περισσότερες από αυτές, εκτός από τις χώρες του κόλπου, οι περισσότερες από αυτές είναι χώρες που έχουν μεγάλο πληθυσμό. Είναι αναδυόμενες χώρες που έχουν τη δικιά τους ανάπτυξη και που όλο και περισσότερο βρίσκονται υπό την πίεση της βιομηχανίας και του τοπικού πληθυσμού, όπως η Αλγερία για παράδειγμα, για να προσφέρουν περισσότερη ενέργεια στον τόπιο πληθυσμό είτε υπέρ της βιομηχανίας, είτε υπέρ του τουρισμού και άρα χρειάζεται, χρειάζονται περισσότερη ενέργεια. Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν, πολύ συγκεκριμένα, ε, πριν από δύο χρόνια δεν συνέβαινε αυτό, τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει μια ε, ενδυνάμει σύγκρουση, διότι τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουν αυτές οι χώρες. Πρέπει να φροντίζουν για περισσότερο συνάλλημα από την Ευρώπη εξάγοντας ενέργεια ή πρέπει την ενέργεια αυτή να την κρατήσουν για τη δικιά τους την ανάπτυξη. Αυτές οι συγκρούσεις που ακόμα είναι υποσκάπτουσες μπορεί να εμφανιστούν πολύ πιο έντονα στο μέλλον στην Αλγερία, στην Αίγυπτο με κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συγκρούσεις. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι Αίγυπτος. Το 2008 πάγωσε η Αίγυπτος κάθε επιπλέον εξαγωγή φυσικού αερίου, όχι μόνο προς τους Ευρωπαίους, αλλά και προς τους γειτονές της, με τους οποίους έχει ε, συμβάσεις Συρία, Ιορδανία και Λίβανο. Πάγωσαν και η Αλγερία από την άλλη μεριά που έχει μια δικιά της ενεργειακή πολιτική του Υπουργού που έφυγε πέρσι, η πολιτική αυτή αντικαταστάθηκε από μια πιο συντηρητική με προσανατολισμό περισσότερες εξαγωγές από τον τωρινό Υπουργό Ενέργειας. Όταν λοιπόν εμείς οι Ευρωπαίοι σκεφτόμαστε ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τον ενεργειακό εφοδιασμό των χωρών αυτών, των προμηθευτών μας. Αυτοί αν έχουν αρκετή ενέργεια. Κάτι πιο τεχνικό, αλλά είναι σημαντικό και αυτό. Είναι το εξή. Ώστε οι χώρες του Νότου που ενδυνάμει μπορούν να μας εξάγουν ενέργεια. Αν θέλουν να καλύψουν και τις δικές τους ανάγκες που είναι αυξανόμενες και ε, τις δικές μας τις αγορές, πρέπει να διασφαλίσουμε ε, μακροπρόθεσμα εφοδιασμό από αυτές. Και προς το παρόν, ξέρουμε ότι το φυσικό αέριο μας καλύπτει εφόσον έχουμε και προσαρμογή των τιμών και μακροχρόνιες συμβάσεις. Το φυσικό αέριο ξέρουμε ότι συνδέεται με το πετρέλαιο όσον αφορά τις τιμές. Ωραία. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και σημεία όπου ξέρουμε ότι βρίσκεται στο υπέδαφος φυσικό αέριο και θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε και αυτό. Και ο λόγος είναι ότι οι διάφοροι διαχειριστές, είτε Σολατράκ ή άλλοι, στις χώρες του Νότου, αλλά και άλλοι, ψάχνουν περισσότερο φυσικό αέριο. Είναι δηλαδή εταιρείε που ασχολούνται και με το πετρέλαιο και με το φυσικό αέριο. Θέλουν και πετρέλαιο και φυσικό αέριο που είναι διατεθειμένες να κάνουν μεγάλες επενδύσεις στην έρευνα για φυσικό αέριο, αλλά θα το κάνουν μόνο αν ξέρουν ότι θα έχουν τα ίδια κέρδη με αυτά που θα είχαν αν κάνανε περισσότερη έρευνα για πετρέλαιο. Φαίνεται ότι μακροπρόθεσμα θα εξακολουθεί να υπάρχει η στενή σχέση ανάμεσα στην τιμή του πετρελαίου και την τιμή του φυσικού αερίου. Όταν δηλαδή θα έχουμε 150 δολάρια το ε, πετρέλαιο, το αντίστοιχο σε φυσικό αέριο θα έχει μια παρόμοια τιμή. Για να μην μπω και μεγαλύτερη, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την μεταφορά. Λέω μακροπρόθεσμα, γιατί πρέπει να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε το μέλλον. Και γι' αυτό λέω ότι οι διάφορες εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να κάνουν μεγάλες επενδύσεις αν δεν ξέρουν ότι θα έχουν μακροχρόνια συμβόλαια. Αν είναι για λίγους μήνες ή λίγα χρόνια δεν τους φτάνει. Φτάνουμε στο τέλος της ανάλυσης αυτής. Και εδώ υπάρχουν κάποιες συστάσεις. Όσον αφορά τον ηλεκτρισμό και την ενεργειακή απόδοση. Οι συστάσεις μας μιλάνε για στήριξη των κέντρων ανασεώσιμων ε, πηγών ενέργειας στις νότιες χώρες. Υπάρχουν οργανισμοί στο Μαρόκο, για παράδειγμα, που μόλις δημιουργήθηκαν, όπως η Εντερέ, που είναι ένα κέντρο για τις ανασεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Τινησία επίσης υπάρχει το ΕΝΕΜΕ Υπάρχει η Εθνική Ένωση Ελέγχου Ενέργειας. Στην Αίγυπτο επίσης έχει δημιουργηθεί ένα Energy Efficiency Agency και λοιπά και λοιπά. Και αλλού και στην Ιορδανία υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Άλλη σύσταση είναι να επεκτείνουμε τον μηχανισμό Έλενα, European Local Energy Assistance που επιτρέπει να στηρίξουμε κοινά σχέδια και να τα επεκτείνουμε στις χώρες νοτίως της Μεσογείου. Ένα Med Έλενα δηλαδή που θα μπορούσε να υποστηρίξει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άλλη σύσταση. Περιφερειακές συνεργασίες. Υπάρχουν στρατηγική σημασία εταιρικέ σχέσεις που μπορούν να γίνουν μέσω των διαφόρων ενεργειακών πόλων. Στο Μαγκρέπ, για παράδειγμα, αντί να έχουν μία, μάλλον αντί να έχουμε ε, πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μία ή την άλλη χώρα, να έχουμε μία πολιτική για έναν πόλο, τις χώρες του Μαγκρέπ, για παράδειγμα τέτοια συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί ώστε να υπάρξει σύγκληση των ρυθμίσεων που καλύπτουν τον τομέα του ηλεκτρισμού. Και να υπάρχει επίσης και σύγκληση και με την ευρωπαϊκή ρύθμιση. Αυτή η ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία θα μας επιτρέψει και πολύ περισσότερο να ενισχύσουμε τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας, γιατί θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε καλύτερα το γεγονός ότι οι ανανόσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι συνεχούς ροής. Κάτι άλλο τώρα. Πυρηνική ενέργεια. Η Αίγυπτος έχει προβλέψει 8 πυρηνικούς σταθμούς. Ξέρω ότι το θέμα είναι βέβαια επίμαχο, αυτό ίσχυε πριν τη Φουκουσίμα. Τώρα αν έχει αλλάξει η Αίγυπτος δεν ξέρω. Κανονικό πρώτο πυρηνικό σταθμό θα έπρεπε να ξεκινήσει το 2019. Θα αλλάξει το πυρηνικό της πρόγραμμα η Αίγυπτος. Δεν ξέρω. Πιθανόν πάντως να πάει προς αυτή την κατεύθυνση η Αίγυπτος. Άλλες χώρες τώρα όπως είναι το Μαρόκο ε, και αυτοί το σκέφτονται. Ας έχουν αρκετό ήλιο. Σκέφτονται 7% της ενέργειάς του το 2030 να παράγεται από πυρηνική ενέργεια. Άρα οι χώρες αυτές νοτίως της Μεσογείου δεν έχουν καταλήψει την ιδέα της πυρηνικής ενέργειας. Γι' αυτό και πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας και να επιμείνουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία και την ασφάλεια. Και να ε, δώσουμε ό,τι συμβουλές ε, χρειάζονται οι χώρες αυτές. Για το φυσικό αέριο τώρα. Έχει άμεση σχέση με αυτά που σας είπα πριν, ε, η σύστασή μας. Τρεις βλέπω εδώ. Διαφοροποίηση στον εφοδιασμό. Και στήριξη, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη, σε προγράμματα τα οποία μας επιτρέπουν τη διαφοροποίηση στον εφοδιασμό μας, ακόμα και αν αυτό γίνει σε βάρος παραδοσιακών προμηθευτών μας όπως είναι η Ρωσία. Υπάρχει τρόπος και είναι ε, ο νότιος ε, διάδρομος Τουρκία από πηγές πιο ανατολικά που να τροφοδοτεί την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη με έναν κλάδο προς την Ελλάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι έτσι καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης χάρη στο σχέδιο αυτό. Το πώς είναι συζητήσιμο. Αυτό όμω που πρέπει να πούμε είναι ότι η απουσία κοινή πολιτικής ενέργειας στην Ευρώπη οι διάφορες χώρες και οι φορείς πάνω ο καθένας προς τη δικιά του κατεύθυνση. Καλό θα ήταν λοιπόν να δημιουργήσουμε μία μονάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία να αποφασίζει με συγκεκριμένη πλειοψηφία που θα καθοριστεί αργότερα ώστε να μπορούμε να έχουμε μία κοινή πολιτική στα θέματα αυτά με μια ενιαία αρχή. Έτσι θα διασφαλίσουμε τον εφοδιασμό. Τώρα εφόσον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πόλιος ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη ρύθμιση είναι καλό. Υπάρχουν πράγματα πολύ ενδιαφέροντα που δεν υπήρχαν πριν. Οπότε τόσο το καλύτερο. Είναι μέτρα τα οποία τα έχουμε σκεφτεί καλά και έχουν διατυπωθεί πολύ καλά στις ρυθμίσεις αυτές. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο πέρα. Γιατί ως επιτοπλίστων, όσα προβλέπονται από την ρύθμιση, μέτρα υποχρεωτικά και αναγκαία, έχουν να κάνουν κυρίως με την επιθυμία να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία προκύπτουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια χώρα, σε πολλές χώρες και έχουν να κάνουν με τη μεταφορά την παραγωγή φυσικού αερίου. Τώρα όμως χρειαζόμαστε ένα νέο πακέτο μέτρων τα οποία να απευθύνονται στο μετά, δηλαδή τι γίνεται εφόσον υπάρχει πρόβλημα με τον εφοδιασμό από χώρες εκτός Ευρώπης. Και επειδή είμαστε πάντα στο θέμα της διασφάλισης του εφοδιασμού, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο αλλά και αναγκαίο οι διαδικασίες λήψης απόφασης για την ε, οικοδόμηση προγραμμάτων, αγωγών, για παράδειγμα, είτε πρόκειται για τους σιδηρόδρομους, είτε πρόκειται για οτιδήποτε. Οι διαδικασίες που έχουμε σήμερα και οι οποίες κρατάνε πάρα πολύ καιρό Χρειαζόμαστε μερικέ φορέ 10 χρόνια για να φτιάξουμε έναν αγωγό. Πρέπει να μειωθούν οι προθεσμίε αυτέ, κατά το ίμιση τουλάχιστον. Αν μπορούσαμε να έχουμε έναν κύκλο για την κατασκευή ενό streamline ή μια άλλη υποδομή. αν μπορούσαμε να φτάσουμε λοιπόν στα 5 χρόνια αντί για τα 10 που έχουμε σήμερα, θα έχουμε κερδίσει πολλά. Είναι απόλυτα λογικό. ήταν ήδη τεράστια πρόοδος. Ίσως μπορούμε να ακολουθήσουμε και τη διαδικασία που δεν ισχύει μόνο στη Γαλλία φαντάζομαι, δήλωση κοινή ωφελία. Οπότε από τη στιγμή που δηλώνεται κοινή ωφελία ένα πρόγραμμα, τότε οι διαδικασίες για την ε, εκτέλεση του έργου αυτού επιταχύνονται και αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους. Τρίτο, α δεν υπάρχει τρίτο, όχι. Αλλά θα έλεγα ότι είναι πολιτικό αν υπάρχει. Και αυτό είναι ότι η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Και κάτι το οποίο με ενοχλεί εμένα στις ε, προσδοκίες που βλέπουμε στα διάφορα ευρωπαϊκά κείμενα είναι ότι περιμένω από τις αγορές να κάνουν τα πάντα. Δεν γίνεται όμως. Όταν μιλάμε για μια στρατηγική, για ένα τόσο λεπτό θέμα όπως είναι η ενέργεια, και όταν μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια για τις υποδομές, ε, δεν νομίζω ότι η αγορά μπορεί να τα κάνει όλα. Και εδώ λοιπόν πιστεύω ότι έχει νόημα η δημιουργία των ένσω των δικτύων αυτών. Βοηθάει βέβαια. Αλλά χρειάζεται και σχεδιασμός και πώς να το πω, κάποιος να παίρνει την απόφαση και να φροντίζει να τηρείται. Τη δεκαετία του 60 του 70 είχαμε το λεγόμενο κομισαριάτ, μια επιτροπή για τα θέματα αυτά. Εντάξει, δεν λέω να ξαναπάμε σε εκείνη την εποχή απαραίτητα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια κεντρική δίκηση που να επιβάλλει κάποιες αποφάσεις. Μήπως δηλαδή χρειαζόμαστε μία αρχή και περισσότερο σχεδιασμό αντί να περιμένουμε την αγορά να καλύψει τα πάντα. Όσον αφορά τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, υπάρχει μια μεταρρύθμιση τιμών, η οποία θα πρέπει να γίνει επίση, Οι τιμέ του ηλεκτρισμού επιδοτούνται, είναι πολύ κάτω από αυτό που θα έπρεπε να ήταν. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η αλήθεια των τιμών, αν θέλουμε να προχωρήσουμε προς ε, υγιή διαχείριση του τομέα και σύγκληση των ε, ενεργειακών πολιτικών ε, των χωρών μέσα στα περιφερειακά σύνολα. συνδέεται με αυτό η πτυχή της ζήτησης, η διαχείριση δηλαδή με βάση την ζήτηση. Σημαίνει αυτό γνώση της ζήτησης και της διαχείρισής της. Oui, enfin, juste, oui, quelques mots sur le, enfin, on a déjà parlé dans des issues. πρόθεση της ε, ενεργειακής ολοκλήρωσης μέσα στο πλαίσιο των χωρών του Νότου της Μεσογείου συχνά είναι δύσκολο γιατί για, λόγω ιστορικών προβλημάτων και δύσκολων πολιτικών σχέσεων ιδιαίτερα στο επίπεδο του Μακρέβα ανάμεσα στο Αλγερία και τους γείτονές της που δεν είναι πλούσιοι Αντίθετα, αυτό που είναι κρίμα είναι να βλέπουμε ότι η Αλγερία που έχει πόρους ε, φυσικού αερίου και ακόμα και αν ε, πάει σιγά σιγά στις εξαγωγές θα μπορούσε για δεκαετίες να προμηθεύει το Μαρόκο και την Τινησία. Αυτό λοιπόν που είναι λυπηρό είναι να βλέπουμε πως το Μαρόκο δεν έχει αναπτυχθεί στο φυσικό αέριο παρά μόνο μέσω του φυσικού αερίου που πληρώνουν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι ε, που όμως προέρχεται από τη Σονατράκ. Πάει από την Αλγερία στο Μαρόκο και την νησί υπάρχει ένα μικρό εμπορικό, μια μικρή εμπορική σύμβαση που αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι περιορισμένο αυτό που θα μπορούσε να αγοράζει την νησί από την Αλγερία. Υπάρχει δηλαδή έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των χωρών αυτών και υπάρχουν δυνατότητες οι οποίες αν λυθούν τα πολιτικά ζητήματα είναι τεράστιες. Στο ΜΑΣΡΕΚ, χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε αυτό το πρόγραμμα, ε, το Master Plan, Το ζήτησε η Ελλάδα και το δέχτηκαν οι χώρες του Μασρέκ να ενισχυθούν οι ενεργειακοί δεσμοί φυσικού αερίου ανάμεσα στι τέσσερι χώρε με άνοιγμα προ την Τουρκία και το Ιράκ. Γιατί αυτέ οι χώρε είναι παρατηρητέ στι ε, συνεδριάσει του εαεμ Η Αίγυπτος ε, έχει παγώσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου και άρα ο στόχος αυτού του master plan που είναι η δημιουργία μιας εκμετάλλευση του αραβικού ε, ε, αγωγού φυσικού αερίου ανάμεσα στη Συρία, την Αίγυπτο και το Λίβανο έχει παγώσει. λειτουργεί κατά μόνο 25% των δυνατοτήτων της. Πάντως υπάρχει ο σταθερός ε, σύνδεσμος και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι εάν τελικά οι πολιτικές εντάσεις ανάμεσα στο Λίβανο και τη Συρία που διαρκούν εδώ και χρόνια ε, επιληθούν. Τελευταία σειρά συστάσεων αφορούν την ενίσχυση της δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειριστεί και να φτιάξει ένα μεσογειακό πρόγραμμα ή προγράμματα. Καταρχήν το ηλιακό μεσογειακό πρόγραμμα να το διαχειριστούμε καταλήλως. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πάει καλά. Υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να γίνουν. Δηλαδή να υπάρξει μια διαχείριση που θα συνδέει τους βασικούς εταίρους που είναι η Κομισιόν, η Γραμματεία της Βαρκελόνης και η Παγκόσμια Τράπεζα. Και έπειτα να ξεκινήσουν αναλύσεις ώστε να μπορέσει να κλείσει αυτό ο, πε, ο περίφημος κρίκος, το MedRing που σημαίνει ταυτόχρονα τεχνικής φύσης και περιβαλλοντικής φύσης αναλύσεις για το πώς θα ξεπεραστεί αυτό το φυσικό εμπόδιο, η θάλασσα δηλαδή. Αυτά. Ζητούμε συγγνώμη γιατί μακρηγορήσαμε παρουσιάζοντας αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Η κυρία Μαντουρέλ. Δεν είναι όμως παρούσα πια. Η κυρία Γκροστέτ. Ε, σε δύο λόγια. Να σας πω ότι η παρουσίαση αυτή ήταν εξαιρετικά ήδη ενδιαφέρουσα. αλλά βλέπουμε πόσο ευαίσθητα είναι όλα αυτά, πόσο ευάλωτα λόγω της, του χαρακτήρα της ε, πολιτικής των χωρών αυτών της Νοτιού Ευρώπης. Και αυτό βασικό νόημα είναι ανεξαρτησία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ενέργεια. Να μην εξαρτώμαστε μόνο από τους άλλους. Ε, σας ευχαριστούμε για την ε, παρατήρηση αυτή και το θέμα δεν είναι μόνο η εξάρτηση από την ε, Ρωσία, είναι και θέμα επενδύσεων. Νομίζω ότι η παρουσίαση έκανε σαφές πόσο ε, πολύπλοκη τεχνολογικά είναι η υπόθεση αυτή. Ας μην ξεχνάμε και πόσο βαθιά είναι η θάλασσα. Όλα μπορεί να φαίνονται πολύ ε, ωραία και πολύ εύκολα, αλλά ε, μέχρι να πραγματοποιηθούν ε, αυτό απαιτεί χρόνο και χρήμα και παραμένουν και κάποια ερωτήματα. Αλλά ναι, θα τα συζητήσουμε αυτά. Η κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της ομάδας μου, ευχαριστώ πάρα πολύ τους προσκεκλημένους μας. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας, για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για τόσα μας εξηγήσατε. Η έκθεσή σας είναι πολύ καλή, πλήρης, ξεκάθαρη. Αναμφίβολα θα αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την Επιτροπή μας. Πολλά θέματα από αυτά που θίξατε με ενδιαφέραν ιδιαίτερα. για παράδειγμα, οι συστάσεις που μας δίνεται στο τέλος, ότι έχει να κάνει με την ενεργειακή απόδοση που πρέπει να είναι ε, προτεραιότητα και για τις χώρες νοτίως της Μεσογείου εξαιτία των δημογραφικών εξελίξεων εκεί και ότι δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι μας ε, για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών κτλ. Αναφερθήκατε επίσης στους μηχανισμούς, Ελένα, είπατε ότι μπορεί να υπάρχει ένα MED Ελένα, Ελένα δηλαδή για τη Μεσόγειο. Είπατε πώς ε, θα διασφαλίσουμε το θέμα της ενέργειας στην Μεσόγειο με ε, παράγοντα και τη διακυβέρνηση κλπ. Θα ήθελα όμως να σας υποβάλω δύο ερωτήσεις για να ικανοποιήσω την περιέργειά μου κυρίως γεωπολιτικά πρώτα απ' όλα. Και μετά θα κάνω και ένα σχόλιο. Πρώτον, για δύο πράγματα που λέτε στην έκθεσή σας. Στα συμπεράσματά σας πρόσεξα ότι αναφέρεστε στο δεύτερο τμήμα και λέτε την εξής πρόταση ότι η απουσία ή η έλλειψη ε, διασυνδέσεων νότου-νότου μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση διασυνδέσεων κάθετων, βορρά-νότου. Εμείς όμως λέμε πάντα ότι η ολοκλήρωση, ολοκληρωση σταθεροτητα είναι πράγματα που θέλουμε για τους εταίρους μας, γιατί αν δεν υπάρχει σταθερότητα στις χώρες εκείνες, κινδυνεύει και ο δικός μας ο εφοδιασμός. Ιστορικά, ξέρουμε ότι η ολοκλήρωση στην Ευρώπη ήταν οικονομική, πολιτική κτλ. Οπότε βλέπω εδώ πέρα ένα, κάτι το παράδοξο στα σχόλιά σας αυτά. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω είναι κάτι σχετικά με την Αλγερία. Λέτε ότι πρέπει να συνεχίσουμε, μάλλον λέτε ότι θα ήταν λάθος να ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις μας με την Αλγερία. Υπάρχουν διασυνδέσεις με το Μαρόκο και με την Τινησία. Μα εσείς είπατε ότι θα ήταν λάθος μια ισχυρή διασύνδεση με την Αλγερία. Για σχολιάστε το και αυτό παρακαλώ. Είπατε επίση ότι το πρόβλημα ε, της Ιβηρικής Χερσονήσου σήμερα είναι ότι δεν έχει πελάτες για το αέριο που θα ήθελε να εισάγει από τη Βόρεια Αφρική. Εμείς όμως ξέρουμε ότι το πρόβλημα στην Ισπανία είναι κυρίως η διασύνδεση με τη Γαλλία που δεν είναι καλή θα μπορούσαμε, αν ήταν καλή η διασύνδεση αυτή, να βοηθήσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη σε περίπτωση προβλήματος με την εισαγωγή φυσικού αερίου που μπορούμε να κάνουμε από τη Βόρεια Αφρική. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλατε παρακαλώ να απαντήσετε. Oui, Enfin, collègue Ναι, βεβαίω ο συνάδελφο θα απαντήσει για το φυσικό αέριο. Όσον αφορά τους ε, οριόντιους ε, συνδέσμους και την αδυναμία τους σε σχέση με τους κάθετους συνδέσμους είναι ε, όντως μια δυναμία. Όταν δούμε τις χώρες Μαγκρέμπη, οι ανταλλαγές, οι οικονομικές μάλλον συναλλαγές ανάμεσα στις χώρες είναι πολύ μικρές. 1,3% είναι μόλις, ενώ το 60% αφορά συναλλαγές με την Ευρώπη. Όσον αφορά λοιπόν τα περιφερειακά σύνολα, νομίζω είναι η πιο αδύναμη ολοκλήρωση που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί. Νομίζω πως η ενίσχυση αυτών των δεσμών θα επέτρεπε να έχουν και πιο ισχυρούς και βιώσιμους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχο πρέπει να είναι η περιφερειακή ευημερία, δηλαδή οι χώρε αυτές να αντιμετωπίζονται σε ένα περιφερειακό σύνολο και άρα κατά συνέπεια το πρόβλημα της Αλγερίας θέλουμε να το χειριστούμε γιατί αυτή είναι η μεγάλη ενεργειακή δύναμη από τι τρει χώρε. Το Μαρόκο δεν έχει καθόλου φυσικό αέριο και ούτε και την Ισία. Έχουμε λοιπόν την τάση να μιλάμε μόνο με την Αλγερία. Ε. Και θα πρέπει να την ξεπεράσουμε κάπως αυτή την τάση. Οι χώρες αυτές φτιάχνουν ισχυρού δεσμούς για το ενεργειακό, στο ενεργειακό επίπεδο και πρέπει να τις στηρίξουμε. Υπάρχει το πρόγραμμα ολοκλήρωσης των μαγρεμπινών ε, αγορών ενέργειας Είχα το προνόμενο το, να ηγούμε του προγράμματος αυτού το οποίο χρηματοδοτεί η Κομισιόν και σταμάτησε κάποια στιγμή γιατί η ευρωπαϊκή στήριξη σταμάτησε. Δεν υπάρχει πλέον δηλαδή τεχνική στήριξη μετά από τον Ιούνιο του 2010, αλλά συνεχίστηκε το πρόγραμμα. Και οι τρεις χώρες εξακολουθούν να μιλάνε για το πρόγραμμα αυτό, για την, για την ε, ολοκλήρωση δηλαδή των τριών μαγκρεμπινών αγορών ε, ε, ενέργειας. Υπάρχει δηλαδή πραγματικό ενδιαφέρον. Τώρα όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Είναι βέβαιο ότι η σύνδεση ανάμεσα στην Ισπανία και στην Γαλλία μπορούν να βελτιωθούν. Στο επίπεδο μάλιστα των ηλεκτρικών συναλλαγών θα γίνει αυτό. Έχουν γίνει οι σχετικές μελέτες ήδη. Για το φυσικό αέριο να σας πω ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό διότι Μέχρι πολύ πρόσφατα η Ισπανία ήταν η χώρα που γνώρισε κατά τη διάρκεια των ετών 80 με 2000 την πιο σημαντική ανάπτυξη προς το φυσικό αέριο με την κατασκευή 12 ε, σταθμών επαναέρωσης, επαναεροποίησης και αλλά εκεί σταματούσε το φυσικό αέριο στην Ισπανία. Δεν υπήρχε δηλαδή αγωγό. Αυτό αλλάζει όμω τώρα, διότι χάρη στο πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υπάρχει, δεκα, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της... περιοχής των Ανατολικ... Ε, Δυτικών Πυρηναίων. Η Ισπανία θα μπορεί να εξάγει προς την Γαλλία και τούμπαλιν. Αυτό θα επιτρέψει στη Γαλλία και σε άλλες χώρες πέρα από τα γαλλικά σύνορα να λαμβάνουν φυσικό αέριο που προέρχεται από την Αλγερία μέσω της Ισπανίας. Αυτό μακροπρόθεσμα είναι πολύ θετικό από στρατηγική άποψη και θα επιτρέψει τόσο στην Ισπανία όσο στην Γαλλία όσο και στην Πορτογαλία να μπορούν να έχουν προσωρινέ ή συγκυριακέ παραδόσεις ανεφοδιασμού αν υπάρχει πρόβλημα σε κάποια από αυτές τις χώρες. Τώρα, το γεγονός ότι η Ισπανία, όπως και η Ιταλία, βρέθηκαν το 2009 και 2010 σε δύσκολη κατάσταση διότι οι συμβάσεις φυσικού αερίου που αγόρασαν ε, ήταν μεγαλύτερες από τη ζήτηση, αυτό είναι κάτι συγκυριακό, δεν είναι κάτι διαρθρωτικό. Για να επανέλθω τώρα στα όσα είπατε, γιατί μιλήσαμε για την ανάγκη επιτάχυσης της διαδικασίας κατασκευής υποδομών και μιλούσα κυρίως για αγωγούς φυσικού αερίου διασυνοριακούς αλλά και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων και μάλιστα σκεφτόμουν ε, τις ε, ενότητες ε, Μεσογείου. Μιλάμε για χώρες οι οποίες είναι κοντά ε, σε επίπεδο ανάπτυξη, Ιταλία και Ισπανία. Αυτό το οποίο όμω είναι εντυπωσιακό είναι ότι η Ισπανία μέσα σε 10-12 χρόνια κατασκεύασε 12 σταθμού επαναεροποίηση, ενώ είχε ήδη τρει και αυτή η κατασκευή έγινε γρήγορα και αποτελεσματικά διότι αυτές οι εγκαταστάσεις είναι κέντρα δραστηριότητας και επέτρεψαν στην Ισπανία να γίνει μεγάλη χώρα στο φυσικό αέριο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ένας από τους σημαντικούς παράγοντες, παράγοντες κλειδί που επέτρεψαν την υλοποίηση των υποδομών ήταν ότι οι επαρχίες της Ισπανίας κατάλαβαν ότι ήταν αναγκαίο να φτιαχτούν αυτοί οι σταθμοί και οι κεντρικές κυβερνήσεις αλλά και οι ιδιώτες είχαν πολύ θετική αντίδραση για την ανάπτυξη αυτών των σταθμών. Ενώ απέναντι οι Ιταλοί, οι Ιταλοί τσακώνονται εδώ και 25-30 χρόνια για να φτιάξουν ε, σταθμούς επαναεροποίησης με μεγάλη, με, χωρίς αποτελέσματα, με τα αντίθετα αποτελέσματα από την Ισπανία. Γιατί η διαδικασία στην Ιταλία δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν τέτοιου είδους υποδομές. Αν μπορούσε δηλαδή να φτιάξει η Ευρώπη ένα σύστημα που να επιτρέπει όταν πρόκειται για υποδομές κλειδιά τέτοιου τύπου και φυσικά μετά υπάρχει το θέμα των πολιτικών αποφάσεων, των ψήφων κτλ. που θα επέτρεπε την επιτάχυση της κατασκευής τέτοιου είδους υποδομών θα ήταν σίγουρα εξαιρετικό, ε, εξαιρετική εξέλιξη για την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Δύο λόγια για τις παρατηρήσεις της ε, κυρίας, ε, την πρώτη σας παρατηρήση. Εδώ μιλώ για φυσικό αέριο, εσείς μιλήσατε για ηλεκτρισμό, θα πρέπει να δείτε με τον Μπερνάρ, ότι... αλλά το πρόβλημα όσον αφορά το φυσικό αέριο είναι ότι το επίπεδο ανεξαρτησίας, μάλλον εξάρτησης από το φυσικό αέριο στο οποίο βρίσκεται η Ευρώπη, δεν δεν είναι επικίνδυνο επειδή εξαντλώνται τα αποθέματα. Το θέμα δεν είναι δηλαδή να βρεθούν πόροι προμήθειας ε, ε, ε, φυσικού αερίου στην Ευρώπη και ούτε και αυτό είναι κανένα δύνατο. Απλώς πρέπει να εξασφαλιστούν από τεχνικής άποψη οι εξωτερικοί μας προμηθευτές μέσω αγωγών φυσικού αερίου του τύπου Ναμπούκο και όχι South Stream, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη, και να και οι χώρες οι οποίες θέλουν να εξάγουν αέριο προς την Ευρώπη να μπορούν και να το κάνουν. Έτσι ώστε η ενεργειακή, ο ενεργειακός ανεφοδιασμός να είναι επαρκής και κυρίως να λαμβάνονται υπόψη οι εσωτερικές ανάγκες γιατί διαφορετικά σε κάποιους μήνες, εβδομάδες ή χρόνια θα έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε εκρήξεις αλλά δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι πολύ σοβαρός προβληματισμός αυτός και ουσιαστικός. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Ε, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε απότομα, διότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μου και δύο υπουργοί μας περιμένουν έξω. Σας ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες ε, αυτές. Ε, περιμένουμε την μελέτη. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. zufrieden. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Μία ώρα έχουμε προβλέψει και θα ήθελα πραγματικά να εκμεταλλευτούμε καλά το χρόνο. Είναι μεγάλη μου χαρά να ε, καλωσορίσω δύο υπουργούς ε, της Ουγγρικής ε, κυβέρνησης. του γνωρίζετε ήδη, είχαμε επανειλημμένα τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί τους. Είναι, είναι λοιπόν παρόντες εδώ σήμερα. Σας καλωσορίζω θερμά. Ε, ποιος από τους δυο σας θα ξεκινήσει. Καλά, δεν θα μάθω ποτέ τα ονόματα. ζητώ συγγνώμη. Μπορείτε να ξεκινήσετε αν το επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχω συνηθίσει να μην προφέρω σωστά το όνομά μου. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ και να σας αναφέρω τότε τις προόδους ε, της Ουγγρικής ε, Προεδρίας κατά τη διάρκεια αυτών των 180 ημερών. ευχαριστήσω ε, όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα αυτής της ε, Επιτροπής που μας βοηθήσατε στα, στις πολύ σημαντικές προκλήσεις που είχαμε πίσω μας. Ε, είδαμε πολύ ταραχμένες εποχές στην Ευρώπη, δεν χρειάζεται να σας τα θυμίσω όλα αυτά. νομίζω ότι όλα τα γεγονότα αυτά ξύπνησαν την Ευρώπη. Πριν δύο μήνες ε, βρέθηκα εδώ στις Βρυξέλλες ε, και ε, ο Ξαβιαρόλε που είναι υπεύθυνο της ομάδας για τα χρηματιστήρια μας είπε ότι η Ευρώπη κοιμότανε. Θα συνοψίσω λοιπόν εγώ την κατάσταση. Ε, τα δάνεια ήταν το υπνοτικό, ο κόσμος ε, τεμπέλιασε. Σίγουρα πάντως υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα. Από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη διάσωση. Ε, αν ανοίξετε την εφημερίδα θα διαβάσετε ένα σωρό ειδήσει ε, σχετικά με την ε, ανικανότητα πληρωμής και άλλα. Η δημοσιονομική σταθερότητα, η χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι σημαντική. Από μόνη της όμως δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας και δεν αυξάνει την ε, παραγωγικότητα δεν ε, δημιουργεί ανάπτυξη. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε την ανταγωνιστικότητα και να φροντίσουμε ένα ε, περιβάλλον φιλικό προς τους επιχειρηματίες. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και πώς μπορούμε να έχουμε ανάκαμψη με νέες θέσεις εργασίας. Δύο πράγματα είναι σημαντικά. Ε, οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερη ενιαία αγορά, λιγότερο κατακαιρματισμένη αγορά από ό,τι έχουμε στην Ευρώπη. Δεύτερον, χρειάζονται λιγότερη γραφειοκρατία. Πρέπει να βοηθήσουμε τις ε, επιχειρήσεις να μειώσουν το ε, γραφειοκρατικό άχθος. Επίσης ε, χρειάζονται ένα ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να απελευθερωθούν οι δυνατότητες ε, καινοτομίας των επιχειρήσεων αυτών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα. Ε, περισσότερη ενιαία αγορά, λιγότερο κατακαιρματισμένη αγορά. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά επιτεύγματα της Ουγγρικής Προεδρίας ήταν η πράξη για την ενιαία αγορά, η Single Market Act, την οποία υιοθετήσαμε τον Μάιο. Αυτή αποτελεί οδικό χάρτη για τον επόμενο 1,5 χρόνο, ε, θέτοντας 12 προτεραιότητες. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες ε, τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά. Οι τρεις πιο σημαντικές είναι οι εξής. Πρώτον, ε, δεν είναι μόνο κατακαιρματισμένη η ενιαία αγορά, αλλά και οι πολιτικές είναι κατακαιρματισμένες ανάμεσα σε διάφορες επιτροπές στο Κοινοβούλιο. Και πολλοί ε, επίτροποι ασχολούνται με το θέμα αυτό. Δεύτερον, έχουμε την πρόκληση Delors. Νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουν αυτό καλά. Όλοι ξέρουν τη γνωστή φράση ότι κανείς δεν πρόκειται να ερωτευτεί την ενιαία αγορά. Χρειαζόμαστε ε, τη στήριξη του κοινού και ε, έχουμε μια προσέγγιση επίλυσης ε, των προβλημάτων στην ενή αγορά και χρησιμοποιούμε πολύ περίεργες φράσεις, ε, σημεία συμφόρησης, ότι είναι ακόμα μητελής Οι απλοί πολίτες δεν καταλαβαίνουν αυτές τις εκφράσεις. Νομίζω ότι αν επικεντρωθούμε στα προβλήματα της ενιαίας αγοράς δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το, το συνολικό πρόβλημα. Χρειαζόμαστε μια ε, οριζόντια στρατηγική και νομίζω ότι η πράξη για την ενιαία αγορά, η Single Market Act, μπορεί να ε, παράσχει ακριβώς μια τέτοια πλατφόρμα και γι' αυτό χαίρομαι που η Ουγγρική Προεδρία κατάφερε να προοδεύσει στο θέμα αυτό, ώστε να έχουμε μία εμβαθμένη και επικαιροποιημένη ενιαγόρα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ενιαγόρα είναι ένα από τα είναι ένα από τα βασικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η ενιαία αγορά οδηγεί στην ε, καινοτομία. διότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην ενιαία αγορά και την καινοτομία, διότι όσο μεγαλύτερη η αγορά τόσο ε, πιο πολύ συμφέρει να επενδύσει κανείς στην καινοτομία. Σκεφτείτε την Ουγγαρία με 10 εκατομμύρια πολίτες, ε, εάν παράγει κανείς κάτι για αυτήν την μικρή αγορά ε, και χρειαστεί να επενδύσει στην καινοτομία, αυτό διαφέρει από το όταν μπορεί κανείς να αναπτύξει κάτι το οποίο θα απευθύνεται σε μια αγορά μισού εκατομμυρίου. Από την άλλη, αν έχουμε και μια επικαιροποιημένη, ε, μια σύγχρονη και ε, ολοκληρωμένη ενιαία αγορά, αυτό θα είναι κίνητρο για την καινοτομία. Υπάρχει λοιπόν άμεση σχέση ανάμεσα στην ε, ενιαία αγορά και στην καινοτομία. Και αυτό είναι ο λόγος που πιστεύω ότι η ίδια η ενιαία αγορά μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της καινοτομίας. Η δήλωση αυτή του Ξαβιέρου λέει ότι η Ευρώπη κοιμόταν, πήρε υπνοτικό. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ επίκαιρη αυτή η φράση. Κοιτάξτε την τελευταία δεκαετία. Η, την καινοτομία την αφήσαμε να ασχολείται με τον εαυτό της. Ε, ενώ χρειαζόμαστε τεράστιες αλλαγές στον τομέα αυτών. Πριν τρεις μήνες ακούσαμε την ε, γνωστή δήλωση ότι για να υπάρξουν θέσεις εργασίας θα πρέπει να είμαστε πιο καινοτόμοι και πιο μορφωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τον υπόλοιπο κόσμο στην καινοτομία και στην εκπαίδευση. Το χρειαζόμαστε αυτό διότι υπάρχουν πολλά κενά. Αν εξετάσουμε το ευρωπαϊκό τοπίο όσον αφορά την καινοτομία σε παγκόσμια κλίμακα, μπορούμε να δούμε τα, τις ελλείψεις που έχουμε σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Ε, ακόμα και οι ε, επενδύσεις ε, δείχνουν το χάσμα αυτό. Η Ιαπωνία επενδύει 1,5% το χρόνο στην έρευνα και την ανάπτυξη και σίγουρα κάθε χρόνο το χάσμα αυτό θα μεγαλώνει και θα βαθαίνει. Έχουμε λοιπόν προσαρμόσει και τις φιλοδοξίες μας. Έχουμε την, ε, το γνωστό φιλόδοξο στόχο του 3% για την έρευνα και την ανάπτυξη και αν κοιτάξετε τα πρόσφατα στοιχεία για τα εθνικά προγράμματα. Ε, κατά μέσο όρο ε, το ποσοστό φτάνει το 2,7-2,8%. Σίγουρα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Υπάρχουν και κάποιες ανισορροπίες αν κοιτάξετε τις δυνατότητες επενδύσεων και ε, έρευνα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης δεν, είναι, δεν υπάρχει ισορροπία όσον αφορά τα δύο φύλλα. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν πολλά βήματα Εάν κοιτάξετε όμως αυτό που υπόθηκε δεν είναι και καινούριο. Ε, χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να πω ότι η Ουγγρική Προεδρία μπόρεσε να κάνει ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά το ενιαίο σύστημα πληρωμών. Τον ε, Μάρτιο δόθηκε το πράσινο φως για κάτι τέτοιο. Στις 10 ε, Δεκεμβρίου επί Βελγικής Προεδρίας είχαμε μία μακρά συνεδρίαση όπου πετύχαμε πολλούς συμβιβασμούς. Δεν μπόρεσε όμως να επιτευχθεί γενικός συμβιβασμός 10 χώρες λοιπόν είπαν ότι θέλουν να υποβάλουν πρόταση για το θέμα αυτό των ε, πληρωμών ε, της ε, συνεργασίας. Τελικά 25 χώρες υπέβαλαν σχετική πρόταση. Στην συνέντευξη τύπου μετά από την απόφαση αυτή είπα πολύ ταπεινά ότι η ιστορία έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό, διότι 50 χρόνια περιμέναμε αυτό το ενιαίο σύστημα. Τώρα ε, κοιτάμε τα εφαρμοστικά μέτρα και ελπίζουμε ότι στις 27 Ιουνίου ε, κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία και για το θέμα αυτό. Το δίπλωμα το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι σημαντικό ε, επειδή ε, είναι κάτι το οποίο θα προσελκύσει ιδιωτική ιδιωτικές ε, επενδύσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε σύντομα το θέμα του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας να το εφαρμόσουμε σύντομα δηλαδή. Στην ε, καινοτομία η βασική μας ε, πολιτική, το βασικό μας καθήκον ήταν να προετοιμάσουμε το δρόμο για ε, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Είχαμε την ενδιάμεση αναθεώρηση του εβδόμου προγράμματος πλασίου και σιγά σιγά κινούμαστε προς το κοινό στρατηγικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ πιο απλό και ολοκληρωμένο. Προβλέπει έτσι πιο καλή χρήση των χρηματικών και άλλων πόρων, ώστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας στην έρευνα και την ανάπτυξη. Προσπαθούμε έτσι να ε, αντιμετωπίσουμε τις ε, κοινωνικές προκλήσεις ε, και να ενισχύσουμε τις ε, επιστήμες, διότι χωρίς αυτές ε, δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτή την ανάπτυξη. Σιγά σιγά λοιπόν βήμα-βήμα προχωράμε. Κινούμαστε προς το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που ήταν βασικό μας καθήκον και λίγα λόγια για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση της Small Business Act της ε, πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις ε, ήταν σημαντικό βήμα. Έχω μάθει ότι κατά καιρού χρειάζονται κάποια βήματα για να ενισχύσουμε τη θέση μας και για να θέσουμε το θέμα υψηλά στην ημερήσια διάταξη. Ε, η Small Business Act σίγουρα είναι ένα από τα βήματα αυτά. Γίνονται εκεί σημαντικά βήματα για τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ απτά αποτελέσματα από τη μείωση των υποχρεώσεων υποβολής λογαριασμών, για παράδειγμα, για τις μικρές οντότητες, για έναν πολύ μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι έτσι έχουμε διευκολύνει την καθημερινή τους δουλειά. Όσον αφορά την πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλε. και αυτή αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εργασίας μας για πρώτη φορά στην ιστορία. Ε, καταφέραμε να ε, συμφωνήσουμε σχετικά με την πολιτική για το διάστημα. Δεν ήταν εύκολο, νομίζω όμως ότι και αυτό ήταν βασικό ε, ε, βήμα προόδου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές για την επικοδομητική συνεργασία μας. Έχω μάθει πολλά κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας. Ε, ένα είναι ότι πάντα υπάρχουν τρεις παράγοντες, ε, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν. Σίγουρα στο Συμβούλιο έχουμε πολλούς περισσότερους ε, διαφορετικούς παράγοντες, έχουμε 27. Ε, το θέμα είναι πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε τις προσπάθειές μας, ε, διότι εάν ένας από όλους αυτούς καθυστερήσει δύο-τρεις εβδομάδες ή ένα μήνα, είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε να εναρμονίσουμε τις εργασίες μας, τις προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την υποστήριξή σας. Μία φράση Νομίζω ότι καταφέραμε ό,τι ήταν δυνατόν να πετύχουμε. Δεν είναι όλα δυνατά, από πολλές απόψεις. Υπάρχουν διάφορες δυσκολίες. Νομίζω όμως ότι η Ουγγρική Προεδρία μπόρεσε να ξυπνήσει την Ευρώπη με πολλούς τρόπους. Ε, το σύνθημά μας ήταν «Ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη» και ελπίζουμε ότι έχει ενισχυθεί η Ευρώπη κατά το σχετικά σύντομο αυτό χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την ε, παρουσίαση σας αυτή, για την ομιλία σας, αλλά και για τα τελευταία σας λόγια. Είναι πράγματι ε, δύσκολη δουλειά στην Ευρώπη, χρειάζεται προσπάθεια, κατανόηση, πειθαρχία από όλους ώστε ε, να μην ε, καθυστερούμε. Αλλά ε, μέχρι τώρα έχουμε λειτουργήσει πολύ καλά. Επόμενος ο μιλητής. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές της Επιτροπής, βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας πω πώς έχουμε προχωρήσει κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής ε, Προεδρίας ε, όσον αφορά τις τεχνολογίες, ε, τεχνολογίες και πληροφορικής. Θα είμαι σύντομος, γραπτός σας έχω υποβάλει τα αποτελέσματα της εργασίας μας. Ο χρόνος τρέχει. Αρχές Ιανουαρίου είχαμε επισκεφτεί την Επιτροπή σας, την Επιτροπή Ήτρε, για να συζητήσουμε τα σχέδια της ε, Ουγγρικής Προεδρίας για το ε, επόμενο εξάμεινο. Ήταν αρκετά απλή η θέση μας. Ε, Βελγική Προεδρία είχε, ετοιμάσει, είχε προετοιμάσει πολύ καλά τα θέματα. Εμείς απλά έπρεπε να τα επαναλάβουμε. Ε, όσον αφορά τον τομέα μας, ε, ε, στρατηγική, ε, εύρος και ασφάλεια ήταν ε, τα, οι τρεις λέξεις κλειδιά για την Ουγγρική Προεδρία. Όσον αφορά την στρατηγική, θέλαμε να εφαρμόσουμε την ψηφιακή ατζέντα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ψηφιακή ατζέντα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Η υιοθέτηση και εφαρμογή της ψηφιακής ατζέντα ε, αποτελεί ε, κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας ε, της Ευρώπης. Ήταν πολύ σημαντικό να συνδυάσουμε τις διάφορες εθνικές στρατηγικές με την ψηφιακή ατζέντα και ακριβώς γι' αυτό στις 27 Μαΐου κάτω το Συμβούλιο για τις Τηλεπικοινωνίες καταφέραμε να προχωρήσουμε. Είχαμε την πρόθεση της ψηφιακής ατζέντα ε, στην ημερήσια διάταξη και είχαν οι υπουργοί τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την κατάσταση στη χώρα τους. Είχαμε δύο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Από τη μία τους στόχους της ψηφιακής ατζέντας και από την άλλη τις σημαντικότερες προτεραιότητες σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Και δεύτερον, τον ε, στόχο ευρυζωνικό πρόσβαση για όλους μέχρι το 2013. Και σήμερα είναι σημαντική ημέρα όσον αφορά την ψηφιακή ατζέντα. Διότι σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες ε, πραγματοποιείται η πρώτη γενική ε, συνέλευση για την ψηφιακή Ευρώπη όπου θα συζητήσουν οι συμμετέχοντες σε την εφαρμογή της ψηφιακής ατζέντας στην Ευρώπη. Δεύτερο σημαντικό θέμα ήταν ε, το θέμα του ε, φάσματος συχνοτήτων. Χρειαζόμαστε μια κοινή στρατηγική συχνοτήτων στην Ευρώπη. θα πρέπει αυτή να αναπτυχθεί ώστε να δημιουργηθούν και νέες δυνατότητες που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Οι συχνότητες και σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο αποτελούν σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό. Είναι σημαντικός πόρος. Οι συχνότητες είναι πόροι ε, χωρίς ε, τους οποίους δεν θα ήταν καθόλου δυνατή η σημερινή κινητή τηλεφωνία, η ευρυζωνική πρόσβαση λοιπά. Το RSPP, το πρόγραμμα για ε, το ραδιοφωνικό φάσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Πριν κάποιους μήνες, ο Μπάρακ Ομπάμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές χώρες θα ε, ε, επιδιώξουν να έχουν ε, μια κοινή ραδιοφωνική στρατηγική. Επειδή είναι τόσο σημαντική στρατηγική αυτό, είναι σημαντικό η Ευρώπη να μην καθυστερήσει στο θέμα αυτό, όσο γίνεται πιο γρήγορα δηλαδή να υιοθετήσει μια κοινή στρατηγική. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Καταφέραμε σχεδόν ε, να πετύχουμε συνένεση όσον αφορά το RSPP. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν ε, σχετικό έγγραφο ε, που στοχεύει σε, στη συνένεση. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μέχρι τέλος της Προεδρίας και θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι και αύριο θα έχουμε τριμερή διάλογο σχετικά με τις ε, συχνότητες. Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κομισιόν και η Προεδρία θα ε, συμμετάσχουν. Όσον αφορά την ασφάλεια, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα στην Ευρώπη, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πάρα πολλοί πολίτες έχουν κινητό τηλέφωνο, έχουν υπολογιστή. Τα δίκτυα συνδέονται μεταξύ τους. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Και έτσι υπάρχει πρόσβαση και σε προσωπικά δεδομένα. Τον τελευταίο καιρό είδαμε αρκετές επιθέσεις σε τέτοια ε, δίκτυα. Είδαμε και κάποια τεχνικά προβλήματα, ε, λόγω των οποίων ε, κάποιες εκατοντάδες πολίτες έχασαν όλα τους τα αρχεία από τη μία μέρα στην άλλη. Συχνά και για πολιτικούς λόγους ε, είχε περιοριστεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ΕΝΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια του Δικτύου, έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Ουγγρική Προεδρία ξεκίνησε τις εργασίες της που αφορούν την ε, ΕΝΙΖΑ σε μια χαοτική κατάσταση όσον αφορά το μέλλον της υπηρεσίας, διότι δεν μπορούσε να προβλέψει κανείς πόσο καιρό θα συνέχιζε η Ενίζα τη δουλειά της. Ε, και βέβαια είναι δύσκολο να δουλέψει κανείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Θέλαμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας καταφέραμε να ε, παρατείνουμε την εντολή της Ενίζα κατά 18 μήνες. Επόμενο σημαντικό θέμα στον τομέα αυτόν είναι ο εξυγχρονισμός της ΕΝΙΖΑ. θα πρέπει να διατυπώσουμε τις μελλοντικέ αρμοδιότητες και να ξεκαθαρίσουμε και το θέμα της χρηματοδότησης. Όσον αφορά την προστασία ε, κρίσιμων υποδομών, ε, στην Ουγγαρία οργανώσαμε ε, σχετική διάσκεψη. Όλα τα κράτη-μέλη εκπροσωπήθηκαν στη διάσκεψη αυτή. καταφέραμε να υιοθετήσουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Έχουμε το σχέδιο δράσης, έχουμε επιβεβαιώσει άλλη μια φορά το ε, σχέδιο δράσης ε, που είχε υποβληθεί. Επίσης όσον αφορά την ε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αυτός ήταν σημαντικός στόχος της Ουγγρικής Προεδρίας. Κοινός μας στόχος είναι στην Ευρώπη να κάνουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ε, προσβάσιμη για όσο γίνεται περισσότερους πολίτες. Βασικότερος στόχος είναι να παρέχονται καλές αξιόπιστες υπηρεσίες ε, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, Θέλαμε να αυξήσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα ε, με τρόπο αποτελεσματικό ως προς το κόστος. Και εδώ καταφέραμε να σημειώσουμε σημαντικές πρόοδους. Όσον αφορά το ε, πρόγραμμα δορυφορικής πλοήγησης, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δορυφορικής Πλοήγησης, κατά διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας είχαμε μια ενδιάμεση αναθεώρηση και έχουμε υιοθετήσει σχετικά συμπέρασματα του Συμβουλίου τον Μάρτιο στον τομέα αυτόν όσον αφορά το σύστημα Galileo. Ετοιμάσαμε ένα σχέδιο ψηφίσματος ε, για το PRS ε, χθες αυτό ε, υιοθετήθηκε από την Κορεπέρ και αν δεν κάνω λάθος ε, και εσείς το συζητήσατε το ε, τέλος Ιουνίου θα έχετε μια σημαντική ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή Ήτρε και θα σας παρακαλούσα να στηρίξετε την πρόταση αυτή. στην αρχή της Ουγγρικής Προεδρίας υποσχεθήκαμε μια καλύτερη, πιο εντατική συνεργασία με το Κοινοβούλιο, ε, να διατηρήσουμε καλύτερο διάλογο με τους ε, βουλευτές ε, και με τα μέλη της Επιτροπής σας. Ελπίζω ότι τα καταφέραμε, το καταφέραμε αυτό. Ελπίζω και εσείς να το νιώθετε αυτό και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα κάποιους Ευρωβουλευτές για την συνεργασία. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής, τον Χέρμπερτ Ρόιλ, ο οποίος ε, έχει ε, συμμετάσχει τόσο ενεργά στις εργασίες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τράουτμαν, την κυρία Δεκαστήγιο, τον ε, Κούναρ Χόκμαρκ, ο οποίος ήταν η εισηγητής σε θέμα που μας ενδιαφέρει και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους Ούγγρους Ευρωβουλευτές με τους οποίους είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αν έχετε ερωτήσεις, ε, βρίσκομαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω όλα αυτά. Συνεργαστήκαμε πολύ ευχαρίστως και με τους δυο σας και με τους συνεργάτες σας. Και με αυτούς ε, που ε, συνεργαστήκαμε πιο εντατικά κατά τη διάρκεια των τριμερών ε, διαλόγων. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία και ήταν πολύ ευχάριστη η συνεργασία αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που ήταν μαζί μας στην Ουγγαρία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Έχω πολλές καλές αναμνήσεις ε, από την επίσκεψη αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχουν οι συνάδελφοι. Η κυρία Τελκαστήγιο πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Ουγγρική Προεδρία πρώτα απ' όλα για τη δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα θέματα τα οποία απασχολούν την Επιτροπή μας ήδη από την αρχή. Δηλαδή και πριν αναλάβουν την Προεδρία. Όταν είχαμε δηλαδή τη δυνατότητα να βρεθούμε μαζί τους στη Βουδαπέστη, θυμάμαι ότι είχαμε μεγάλη ευκολία να συζητάμε μαζί τους και οι συζητήσεις μας ήταν ιδιαίτερα καρποφόρες. Τώρα φεύγει μια προεδρία και μπαίνει μια άλλη. Κάθε έξι μήνες έτσι γίνεται. Και ένα από τα πράγματα που συμβαίνει κάθε φορά και το λέω από προσωπική εμπειρία, επειδή κάποτε και εγώ στη θέση που είσαστε εσείς τώρα, η κυβέρνηση γνωρίζει τι θέλει το κοινοβούλιο. Οι κυβερνήσεις είναι συνηθισμένες να συνεδριάζουν με την Επιτροπή βέβαια περισσότερο. Οπότε αυτά τα οποία λέει το Κοινοβούλιο είναι κάπως το περιθώριο. Όταν βέβαια ε, παίρνουν την Προεδρία οι κυβερνήσεις ενημερώνονται και τότε καταλαβαίνουν ότι υπάρχει και το Κοινοβούλιο και έχει και αυτό κάποιες ε, απαιτήσει και τότε αποκτάει κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε το κοινοβούλιο μας κερδίζει κάθε φορά που σταματάει μια προεδρία ξέρουμε ότι έχουμε ένα νέο φίλο στο Συμβούλιο, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία κατά την εξάμεινη προεδρία κάθε χώρας να γνωριζόμαστε καλύτερα με τους υπουργούς και με τις κυβερνήσεις. Σας ζητάω λοιπόν και για τα θέματα τα οποία βρίσκονται ακόμα σε κρεμότητα, αλλά και για θέματα που έχουν να κάνουν ε, με το ραδιοφάσμα και για άλλα θέματα σημαντικά, μεγάλα, που θα καλύψουν τις δραστηριότητες σας την επόμενη χρονιά, θέματα έρευνας κυρίως, μην ξεχνάτε τις φιλοδοξίες του Κοινοβουλίου. Και θα σας πω δύο πράγματα ακόμα. Σας παρακαλώ. Εμψυχώνετε τους συναδέρφους σας στο Συμβούλιο από τις άλλες χώρες να κάνουν και αυτοί προσπάθειες, γιατί οι γραμμές στον προπολογισμό για τα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα, ίτερ, Γαλιλαίος κλπ, πρέπει να είναι ειδικέ γραμμές και να μην εμπίπτουν στο γενικό προπολογισμό του προγράμματος πλαίσιο, γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει να πετύχει τους στόχους του το ίδιο το πρόγραμμα πλαίσιο. Δεύτερον, ή δυνατόν προσπαθήστε να αυξηθεί ουσιαστικά 3% να φτάσουμε ή δυνατόν του ΕΠ, όπως έχει ήδη πει το Συμβούλιο της Βαρκελόνης το 2001, αλλά δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι όταν στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε είχαν μεγάλη ύφεση, διπλασίασαν παρόλα αυτά τον προπολογισμό τους για την έρευνα, γιατί ήξεραν ότι η έρευνα θα μπορούσε να τους βοηθήσει να βγουν από την ύφεση πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και στη συνέχεια να γίνουν αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή πρώτη δύναμη στον κόσμο. Αυτό λοιπόν επιθυμούμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασιζόμαστε σε εσά να μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαντουρέλη τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τους δύο υπουργούς που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Και τους ευχαριστώ και για τη δουλειά τους. Έχω κάποιες ερωτήσεις, παρακαλώ. Γιατί στα θέματα της έρευνας εσείς δείξατε δύο σημαντικά ε, ζητήματα. Είναι η απλοποίηση η αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαίσιο. Έχουμε εδώ δύο εισηγητές, δεν θα πω στις λεπτομέρειες, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι οι εκθέσεις τους είναι πάρα πολύ καλές, με πολύ σημαντικά συμπεράσματα προς εφαρμογή. Οπότε, βάσει αυτού, θα ήθελα να γνωρίζω η Προεδρία σας τι έκανε ώστε η Επιτροπή να κάνει πράξη όλα αυτά τα συμπεράσματα, τα τόσο σημαντικά στο οποία καταλήξαμε. Μερικά μπορούν άμεσα να τεθούν σε εφαρμογή, αλλά πρέπει να περιμένουν περισσότερο. Θέλω επίσης να αναφερθώ και εγώ στο 3%. Συμφωνούμε ότι για την οικονομική ανάκαμψη, για να υπάρξει δηλαδή οικονομική ανάπτυξη, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, να έχουμε θέσεις απασχόλησης, ε, ε, εκπαίδευση κατά της κτλ. Αυτός ο στόχος, ο στόχος της Βαρκελόνης, που ήταν στόχος για το 2010, αλλά τώρα έχει πάει για το 2020, εσείς είπατε ότι πρέπει να πάρουμε πολλά μέτρα. Εσείς τι κάνατε, πού πετύχατε σε αυτό, πού δεν πετύχατε, τι μένει, τι αφήνετε δηλαδή για την επόμενη προεδρία σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Αναφερθήκατε επίσης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αναθεώρηση του Small Business Act, SMEs ε, Envoys, τους εκπροσώπους δηλαδή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι μία πρόοδος υπέρ της αντιγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πώς θα πετύχουμε την συνέχεια των πολιτικών, εσείς δηλαδή ποιο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι το επόμενο βήμα μας. Και τέλος, τέλος μην ξεχάσω και τον άλλον υπουργό, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πάλι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχω εδώ ένα κατάλογο με τις πρόδους που έχουν επιτευχθεί, τα ψηφιακά κλπ. Η παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο διαδίκτυο όμως είναι κάτι που έχει πάει λιγότερο καλά. Μπορείτε να μας μιλήσετε περισσότερο γι' αυτό και τι προτείνεται να κάνει η επόμενη Προεδρία από αυτού. Ευχαριστώ. Καβάγιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την Ουγγρική Προεδρία, για την εξαιρετική της εργασία εν Θα ήθελα ωστόσο να τονίσω το εξή. Ήμουν εισηγήτρια για την έκθεση απλοποίηση, απλοποίηση του προγράμματο έρευνα και κοινοτομία και η Ουγγρική Προεδρία έχει παρακολουθήσει το θέμα και την εφαρμογή της εφαρμογή πολύ στενά, σε υψηλό επίπεδο. δημιουργώντας μια άτυπη υποομάδα υπουργών εντός του Συμβουλίου με προεδρία την ίδια την Προεδρία και αυτό έχει συνεργαστεί αυτή η ομάδα πολύ στενά μαζί μας και με την Κομισιόν και ήταν πολύ σημαντική βοήθεια για παράδειγμα για τη δουλειά για τον χρηματοπιστωτικό κανονισμό με τον οποίο ακόμα ασχολούμαστε και ελπίζουμε ότι θα περιληφθεί εκεί θα περιληφθούν εκεί όλες οι αλλαγές που χρειαζόμαστε, ώστε να είμαστε βέβαιοι πως η απλοποίηση των δημοσιονομικών και διοικητικών κανόνων για τα επόμενα ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα καινοτομία θα γίνουν. Και η Ουγγρική Προεδρία έχει προσιλωθεί. Ελπίζουμε ότι θα είστε και σύμμαχό μας σύμμαχός μας για ένα πρόγραμμα πλαίσιο το οποίο θα είναι καταλήλως πρικισμένο. Ο συνάδελφος Κιούρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ε, κυρίους Υπουργούς για την παρουσία του στη σημερινή μας συνεδρίαση. Συμφωνώ με τους συναδέρφους μου ε, ότι η, Ευρωπαϊ... η Ουγγρική Προεδρία βρισκόταν πολύ κοντά στο Κοινοβούλιο. Δεν μας παρουσιάσατε μόνο το πρόγραμμα σας στην αρχή, αλλά και στο τέλος της Προεδρίας σας έχετε το θάρρος να έρθετε εδώ στο Κοινοβούλιο και να λογοδοτήσετε. Αυτό σίγουρα είναι θετικό. Από την άλλη, η Ουγγρική Προεδρία δεν είχε και να φοβηθεί τίποτα κατά την λογοδότηση μετά από το εξάμεινο αυτό. Διότι ο Υπουργό Σεφαρβέη είχε δίκιο. Ήταν ε, δύσκολες εποχές, αλλά η Προεδρία τα κατάφερε. Το πρόγραμμα της Προεδρίας δεν διαμορφώνεται από μια κυβέρνηση, αλλά από την ίδια τη ζωή. Και είδαμε κάποια αναπάντεχα θέματα κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, όπως ήταν η, η κρίση. Δεν ήταν όμως ε, αυτό το θέμα μας σήμερα. Ε, παρά την, ε, παρότι υπήρχε στην ημέρησια διάταξη η διαχείριση των ε, κρίσεων, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και μέσω μακροπρόθεσμα και η απάντηση που θα πρέπει να δοθεί στην κρίση παρόλα αυτά ε, είχαμε και θέματα τα οποία δεν ε, ήταν καθαρά διαχείριση κρίσεων στην ημερήσια διάταξη. Η Ουγγρική Προεδρία έχει κάνει πολλά και έχει θέσει τις κατευθύνσεις για το μέλλον. Ένα ερώτημα συνδέεται με τα θέματα αυτά, έχει να κάνει και με το μέλλον. Έτσι είναι η ζωή, η μία προεδρία φεύγει, η άλλη έρχεται. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με την επικοινωνία και με την ε, πολιτική του ραδιαφωνικού φάσματος. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα της Ουγγρικής Προεδρίας. Στο μέλλον, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την εφαρμογή της πολιτικής, πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε την εφαρμογή της πολιτικής αυτής υπό το φως ε, ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν τρίτες χώρες ως γειτονικές χώρες. Το Κοινοβούλιο έχει υποβάλει την ε, πρότασή του και σίγουρα η Πολωνική Προεδρία θα έχει να κάνει πολλή δουλειά το θέμα αυτό. Η ερώτησή μου όμως είναι εσείς πώς βλέπετε τις δυνατότητες. Η άλλη μου ερώτηση έχει να κάνει με την έρευνα και την ανάπτυξη. Η ενδιάμεση αναθεώρηση του εβδόμου προγράμματος πλαισίου πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Ε, είδαμε όμως ότι δεν ε, έγινε πολύ καλή απορρόφηση των πόρων ε, από όλες τις χώρες. Και είπαν ότι δεν υπάρχει απαραίτητη υποδομή εσείς ε, κύριε Υπουργέ, ε, πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσουν και αυτές ε, οι χώρες χωρίς την απαραίτητη υποδομή να μπορέσουν να φτάσουν σε επίπεδα αριστείας. Επίσης, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε η έρευνα και η ανάπτυξη να μπορέσει να λάβει δικούς τους αποκλειστικούς πόρους. Ευχαριστώ. συγχαρώ και εγώ όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές την Ουγγρική Προεδρία. Η ερώτησή μου είναι κάπως πιο τεχνική. Η Ουγγρική Προεδρία έκλεισε την πρώτη Τρόικα, Ισπανία, Βέλγιο, ε, Ουγγαρία με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Για εσάς... Αυτή η τρόικα ήταν ενδιαφέρουσα, τη χρησιμοποίησατε για θέματα τα οποία είναι μέσα πρόθεσμα, που ξεπερνούν πάντα δηλαδή ε, τους έξι μήνες της, προ, της, της Προεδρίας και η ομάδα του ότι ήταν χρήσιμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω πέντε λεπτά σε καθέναν από τους υπουργούς για να απαντήσουν. Θα ξεκινήσετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πολλές ερωτήσεις και ελπίζω να ήμασταν μια προεδρία φιλική απέναντι στο Κοινοβούλιο. Τουλάχιστον αυτή ήταν ε, η πρόθεσή μας. Και ελπίζω να τα καταφέραμε. Αν τα καταφέραμε, το στο καλύτερο. Να απαντήσω όσον αφορά το 3%. Γιατί πολύ με ρωτήσατε γι' αυτό. Όντω, υπήρξε αυτός ο φιλόδοξος στόχος. Και τι σημαίνει. Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και επενδύσεις και συμμετοχή. Επενδύσει τι σημαίνει. Σημαίνει ότι περισσότερε επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία. Και γι' αυτό είπα ότι χρειαζόμαστε και δέσμευση. Δέσμευση από την βιομηχανία. Είμαι πεπισμένο ότι η καινοτομία είναι κάτι που έχει να κάνει άμεσα με τη βιομηχανία. Τις ξέρουμε τις ιστορίες από το Silicon Valley, όλοι τις ακούμε. Ξέρουμε το, για τον κάρεσα και τον περίφημο τύπο, ο, ο οποίος είχε μια καταπληκτική ιδέα, έγινε ε, εφοπλιστής και μετά τι έγινε κάτι στο Google. Αυτή είναι η ιστορία. Η καινοτομία και η έρευνα είναι πράγματα τα οποία γίνονται από τους διάφορους ερευνητές. Χρειαζόμαστε λοιπόν και την δέσμευση της βιομηχανίας. Και όταν λέμε ότι πρέπει να επενδύσει και η βιομηχανία, άρα πρέπει να φτιάξουμε το κατάλληλο περιβάλλον για αυτή, το κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον. Άρα χρειαζόμαστε επενδύσεις φυσικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο με δημόσια χρήματα, τα κράτη-μέλη, την Ευρώπη κτλ. Αλλά συγχρόνως πρέπει να δημιουργήσουμε και το κατάλληλο πλαίσιο για τη βιομηχανία. Γιατί η καινοτομία είναι κάτι που όλο και περισσότερο έχει να κάνει με τη βιομηχανία. Αν συμφωνήσουμε με αυτό ω σημείο εκκίνησης, τότε δεσμεύεται και η βιομηχανία. Το τρίτο λοιπόν είναι η συμμετοχή. Και εδώ έρχομαι και σε αυτό που με ρωτήσατε, τι είναι για μένα involvement, συμμετοχή, είναι κάθε ενδιαφερόμενου, κάθε χώρας, κάθε μετόχου, κάθε θεσμικού οργάνου. Όλοι πρέπει να βάλουν μαζί τις προσπάθειές τους. Και αυτό εξάλλου είναι και το αποτέλεσμα της ε, προσωρινής μας έκθεσης. Υπήρχαν κάποιοι εκπρόσωποι με τους οποίους συζητήσαμε ξανά και ξανά και στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Οργανώσαμε και ένα τύπο γεύμα για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα. Καλέσαμε τρεις επιτρόπους, ρεκόρ, ε, παγκόσμιο ρεκόρ, τρεις επιτρόπους είχαμε στο γεύμα αυτό. Χαν, Κος και Μεργαν Κουίν. Και συζητήσαμε και με τους τρεις πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας. Η ερώτηση βέβαια ήταν τι θα γίνει με τις χώρες που υποεκπροσωπούνται. Συζητήσαμε το τι λείπει και καταλάβαμε ότι αυτό που λείπει είναι η βασική υποδομή. Άρα χρειάζεται ενίσχυση στις υποδομές. Ο Επίτροπος υποσχέθηκε ότι θα το ερευνήσει και θα επανέλθει το Σεπτέμβριο. 3% λοιπόν, ακούγεται καλά, αυτό που χρειαζόμαστε είναι επενδύσεις και από το δημόσιο όπως είπαμε, χρειαζόμαστε δέσμευση από πλευρά τη βιομηχανίας και για να υπάρξει αυτή πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο, άρα ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τέλος χρειάζεται συμμετοχή Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε να συμμετέχουν χώρες, περιφέρειες κλπ. κλπ ώστε να συμμετέχουν όλοι στην προσπάθεια αυτή. Έρχομαι στο άλλο τώρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Small Business Act. Πάντα γίνεται ερώτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάντα είναι στην ημερήσια διάταξη. Αλλά εμείς έχουμε στο μυαλό μας κάποιες αλλαγές σε σχέση με το πώς βλέπουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποτέ καμία κυβέρνηση δεν υπάρχει και δεν έχω δει που να μην αγαπάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε πραγματικά. Ξέρετε, ο Σούμερ Χέρτ, Βρετανός ε, οικονομολόγος, ε, ήταν που είχε πει «Small is beautiful», το μικρό είναι ωραίο. Ναι, αλλά το να γίνεται ο μικρός μεγάλος και δυνατός, αυτό είναι ακόμα πιο όμορφο θα έλεγα εγώ. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν όλο και περισσότερο ανταγωνιστικές. Χρειάζεται μια στρατηγική, γιατί πολλοί φορές το σκέφτομαι αυτό, ναι τι ωραίες που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν φτάνει το να τις αγαπάμε. Πρέπει να τις βοηθήσουμε να αναπτυχθούν. Άρα με τις κατάλληλες πολιτικές που θα αναπτύξουμε. Οπότε οι διάφορες ιδέες που ακούγονται είναι σημαντικές. Οι μικρομισές επιχειρήσεις τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Όχι το ότι είναι μικρές, αλλά το ότι είναι μόνες, μοναχικές. Δεν ακούγεται η φωνή τους. Τον υπάρχει λοιπόν ένας, ε, κάποια εκπροσώπησή τους είναι θετικό και χαίρομαι που θα υπάρχει ένας απεσταλμένος σε κάθε χώρα ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απλοποίηση τώρα. Είναι δύσκολη δουλειά. Και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας υπέρ της απλοποίησης. Σε ένα βαθμό είναι διοικητικό ζήτημα, αλλά από την άλλη μεριά είναι και πολιτικό θέμα. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Άρα είναι πολύ καλό όταν συμμετέχει και το ψηλό πολιτικό επίπεδο. Και έτσι έρχομαι και στην τελευταία ερώτηση για την προσέγγιση. Στην απλοποίηση είχαμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των τριών προεδριών της Γαλλικής, της Βελγικής, της Ουγγρικής. Και όσον αφορά ε, την πλήρανση ε, του πληθυσμού με υγεία. Και εκεί είχαμε καλή συνεργασία. Τώρα είναι όμως το τι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η Προεδρία είναι μια διαδικασία από την οποία μαθαίνουμε. Κανείς δεν ήταν στην ακριβώς ίδια θέση, οπότε κάθε φορά μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε, μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας πολλά. Και κάτι προσωπικό που θα σας πω τώρα είναι ότι ακριβώς επειδή συνεργαζόμαστε με την Ισπανική και τη Βελγική Προεδρία και τους Υπουργούς, αν έχουμε κάτι να ρωτήσουμε, μπορούμε να συνεργαστούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, κάναμε μια δήλωση για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους των περιφερειών και τα κλάστερς για την καινοτομία. Ο Βέλγος υπουργό και ο Ισπανός υπουργό εκπροσωπή του των ήταν εκεί. Και είπαμε ότι συνεργαζόμαστε εκεί απέναντι στο κοινό, αλλά και για διάφορα ειδικά προγράμματα, πάνω σε διάφορα ειδικά προγράμματα και σχέδια. Και αυτή τη διαδικασία θα τη συνεχίσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δόθηκε ευκαιρία να αποτελέσω μέρος αυτού του τρίου, αυτής της τριάδας και ελπίζω ότι η ίδια καλή συνεργασία θα υπάρξει και με την επερχόμενη Προεδρία, την Πολωνική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την παρουσία τους στο διαδίκτυο το γεγονός ότι στον σημερινό κόσμο, στη σημερινή Ευρώπη, μία επιχείρηση μπορεί να εμφανίζεται στο διαδίκτυο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι εάν δεν έχει κανείς παρουσία στο διαδίκτυο, τότε αυτό σίγουρα είναι μειονέκτημα όσον αφορά τον ανταγωνισμό σε σχέση με τους άλλους. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμείνουμε στους στόχους της ψηφιακής ατζέντα και να τηρήσουμε τις προθεσμίες, διότι στον τομέα αυτών θα μπορέσουμε έτσι να πετύχουμε σημαντική πρόοδο. Θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω το παράδειγμα της Ουγγαρίας τον τελευταίο καιρό. Ε, έχει μειωθεί η διεκπαιρέωση των... Έχει μειωθεί η γραφειοκρατία όσον αφορά την καταχώρηση νέων ε, domain names, νέων ε, ονομασιών στο διαδίκτυο. Θέλουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να εφαρμόσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τους στόχους της ψηφιακής ατζέντα. Όσον αφορά το πολιτικό πρόγραμμα με τις ραδιοφωνικές συχνότητες. Το γεγονός ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία συνορεύουν με τρίτες χώρες. Αυτό σίγουρα είναι ε, θεμητό ερώτημα και θα πρέπει να εξεταστούν οι πρακτικές πτυχές. Ε, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας μας ασχοληθήκαμε με τις πτυχές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Συχνοτήτων θα πρέπει να υιοθετηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο φάκελος έχει υποβληθεί και Ε, θέλουμε, προτείνουμε πρακτικό συντονισμό των ραδιοφωνικών συχνοτήτων. η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προετοιμαστεί καλά για την διεθνή διάσκεψη ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Η καλή συνεργασία της Τρόικα Όσον αφορά την καλή συνεργασία της ε, Τρόικας, ε, κάτι που ρώτησε ένας ε, Ευρωβουλευτή, να έχει λειτουργήσει πολύ καλά και με τους Βέλγους συνεργαστήκαμε καλά, είχαν προετοιμάσει πολύ καλά τα θέματα που, αναλάβα, τα θέματα που αναλάβαμε και τώρα στο τέλος της Τρόικας αυτής, αλλά βρισκόμαστε σε επαφή και με την συνεργαζόμαστε στενά και με την ε, Πολωνική Προεδρία που είναι η πρώτη της επόμενης ε, τριάδας προεδριών. Μέχρι τέλη Ιουνίου θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά. Αύριο, για παράδειγμα, έχουμε τριμερή διάλογο σχετικά με την ε, πολιτική των ραδιοσυχνοτήτων όπου έχει προσκληθεί και η Πολωνική Προεδρία να συμμετάσχει. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας να σας ευχαριστήσω και πάλι. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω αυτά. Σας παρακαλώ να ε, μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας και σε όλους τους συνεργάτες σας ε, που μας βοήθησαν. Ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναβρεθούμε. Το σημαντικότερο είναι ίσως η ελπίδα μας ότι πιστεύουμε ότι έχουμε ένα νέο φίλο στο Συμβούλιο. Διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα ο καθένας που βοηθάει να λυθούν γρήγορα και σοφά τα ευρωπαϊκά προβλήματα ε, είναι φίλος ε, και σημειώνω και αυτό που είπατε εσείς για την θετική οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Καταρχήν θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε θετικά την ε, οικονομία. αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο